Καλό απόγευμα αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Αρχίζουμε λοιπόν τη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Έχουμε σήμερα μαζί μας τον κύριο Πέτερ Ζίγκα, ο οποίος είναι Υπουργός Οικονομίας της Ουραγικής Δημοκρατίας. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ που ήρθατε. Μάλλον επιτρέψτε μου πρώτα απ' όλα να δώσω κάποιες πληροφορίες και ζητώ συγγνώμη που ε, σας καθυστερούμε, αλλά αυτή είναι η ε, διαδικασία. Πρέπει να δώσουμε κάποιες ε, λεπτομέρειες. Πρώτα απ' όλα, εάν δεν υπάρχουν άλλα ε, σχόλια, μπορούμε να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη χωρίς ε, ε, κάποιες τροποποίησεις. Έχουμε συνεδρίαση τριών μισών ημερών μέχρι δηλαδή αύριο στις, 8, συγγνώμη, στις 6 και μισή το απόγευμα. Δεν βλέπω να υπάρχουν σχόλια, επομένως εγκρίνεται. Τώρα, όσον αφορά την σήμανση ενεργειακής ε, απόδοσης, αυτό το θέμα... Αυτό το θέμα ε, επιστράφει στην ε, ε, δική μας Επιτροπή Ήτρε έτσι ώστε να ξεκινήσουν οι συζητήσεις σε επίπεδο τριμερούς διαλόγου υπό τον εισηγητή. και ο πρόεδρος της Επιτροπής επίσης ε, ε, θα ε, συμπεριληφθεί καθώς επίσης και οι σκιώδεις εισηγητές στον τριμερή διάλογο. Ο κύριος Ταμπουράνο θα είναι βεβαίως επικεφαλής της ομάδας διαπραγμάτευσης όπως σας είπα μαζί με τους σκιώδεις εισηγητές. Δεύτερο ζήτημα το οποίο θέλω να σας αναφέρω η απαλλαγή προϋπολογισμού είτε 2014. Η Επιτροπή Ελέγχου του ΕΠ του προϋπολογισμού ε, θα έχει μια συζήτηση και ανταλλαγή απόψε με τον Επιτρόπο Κανιέτε όσον αφορά τη διαδικασία απαλλαγής 2004 για το ΙΤΕΡ και αυτό θα λάβει χώρα την 14η Ιουλίου στις 9 το πρωί όλα τα μέλη της Επιτροπής Ήτρε και αυτό είναι πολύ σημαντικό και το σημειώνω, όλα τα μέλη ε, καλούνται ε, να παραστούν σε αυτήν την ε, συζήτηση. Βεβαίως μπορούμε να είμαστε παρόντες σε οποιαδήποτε επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου θέλουμε μπορούμε να πάμε και να είμαστε παρόντες. Αλλά σήμερα αυτή τη φορά το τονίζω διότι η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού ε, μας έχει αποστείλει μια ειδική πρόσκληση, ε, διότι είμαστε υπεύθυνοι κατά κάποιο τρόπο για το ίτερ. Επαναλαμβάνω λοιπόν αυτή η συνεδρίαση θα λάβει χώρα την 5η 14 Ιουλίου 9 η ώρα το πρωί και παρακαλώ όλα τα μέλη να είναι παρόντα. Και αν σας ενδιαφέρει το θέμα που σας ενδιαφέρει σίγουρα και αν θέλετε να ακούσετε τους συναδέλφους από την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού καθώς επίσης ε, και να συμμετάσχετε, να δώσετε την αποψή σας για αυτή τη συζήτηση, ε, εδώ ε, θα πρέπει να είσαστε παρόντες λοιπόν 14 Ιουλίου. Αυτά ήταν τα σχόλια που ήθελα να κάνω και επομένως μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 3 της ημερησίας διατάξεως. Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επίσκεψη του κυρίου Πέτερ Ζίγκα, Υπουργού Οικονομίας της Σλοβακίας. Για μία ακόμα φορά σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Είναι η πρώτη συνεδρία σας Επιτροπής Ήτρε μετά την ανάληψη της Προεδρίας σας ε, την 1η Ιουλίου και επομένως σας έχουμε αμέσως ε, άμα τη αναλήψη των καθηκόντων σας. Ο κύριος Σαζίκα, ο οποίος ηρίστον παρόδο είναι και δόκτωρ φιλοσοφίας, ασχολείται με θέματα οικονομίας, θέματα μικρομεσαίων ε, επιχειρήσεων και θα ασχοληθεί με διάφορα θέματα τη διάρκεια της Προεδρίας από ό,τι μας έχει πει, κυρίως δε όσον αφορά το πλαίσιο ε, για την σήμανση της ενεργής απόδοσης, όσον αφορά τα στατιστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά το φυσικό αέριο και τις τιμές του, ε, του, του ηλεκτρικού. Επίσης, ε, θα, να σας πω ότι τον Οκτώβρη θα ξεκινήσει ο διάλογος όσον αφορά της διασφά, τη διασφάλιση της ε, ε, ασφάλειας του ανεφοδιασμού όσον αφορά το ε, αέριο. Επίσης θα συζητηθεί και ο μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις διακυβερνητικές συμφωνίες καθώς επίσης και τα μη δεσμευτικά εργαλεία και συμφωνίες μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων χωρών όσον αφορά τον τομέα της ενέργειας. Έχουμε προβλέψει να σας πω 90 λεπτά για αυτήν την ε, συζήτηση. Στρέφουμε λοιπόν προς εσάς, κύριε Υπουργέ, ε, και θα ξεκινήσουμε αυτήν την ε, συζήτηση με τη δική σας παρέμβαση. Έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ για τα πολύ καλά σας λόγια, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι εδώ για να σας παρουσιάσω το πρόγραμμα της πρώτης Σλοβακικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά από 12 χρόνια συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Σλοβακία έχει την τιμή να ηγείται το Συμβουλίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωρίζουμε πόσο σημαντικέ είναι οι εξαιρετικέ σχέσει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είμαστε εκτεθειμένοι να εργαστούμε μαζί σα σε όλου του σημαντικού φακέλου που εξετάζονται αυτή τη στιγμή και αυτή και οι υπόλοιποι θα παρουσιαστούν στο εγγύ μέλλον. Σήμερα θα ήθελα να σα παρουσιάσω τι γενικέ προτεραιότητε τη Λογική Προεδρία και μετά ορισμένα επιμέρου ζητήματα στον τομέα τη ενέργεια και τη ανταγωνιστικότητα. Αυτέ είναι οι κύριε προτεραιότητε, οι δικέ μου ως Υπουργού Οικονομία τη Λογική Δημοκρατία. Οι συνάδελφοί μου, υπουργοί αρμόδιοι για ζητήματα τηλεπικοινωνιών, παιδείας και έρευνα, θα σας ενημερώσουν για τις προτεραιότητες ε, του ε, σχετικού θεματολογίου τηλεπικοινωνιών και έρευνα ε, στη συνέχεια σήμερα και αύριο. Η Σλοβακία αναλαμβάνει τη θέση τη ε, Προεδρία σε πολύ δύσκολου καιρού, αντιμετωπίζοντα και εσωτερικέ και εξωτερικέ προκλήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόσφατη ψήφο και το δημοψήφισμα στο ΕΒ Βασίλειο δείχνουν ότι έχει υπονομευθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να ανακτήσει αυτή την εμπιστοσύνη η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και να επικεντρωθεί σε λύσεις που θα δίνουν μακρόπνοη προοπτική στο ευρωπαϊκό εγχείρημα. Και αυτό σκοπεύουμε και εμείς να κάνουμε προκειμένου να περιορίσουμε και να άρουμε τα εφιστάμενα εμπόδια μεταξύ των μελών. Θέλουμε λοιπόν να είμαστε ρεαλιστές, να ε, ξεπεράσουμε τον κατακαιρματισμό και να θέσουμε ως σημείο εστίαση στον άνθρωπο. Για να επιτύχουμε αυτού του ε, στόχου, έχουμε αποφασίσει να επικεντρωθούμε σε τέσσερι βασικέ αρχέ. Ενίσχυση τη ευρωπαϊκή οικονομία, εξυγχρονισμό και διεύρυνση τη ενιαία αγορά, σε τομεί όπω η ενέργεια και η ψηφική οικονομία ε, η προώθηση της βιώσιμης μετανάστευσης και πολιτικής ασύλου και ενίσχυση της ε, συνολικής δέσμευσης ε, για την Ευρώπη. Πιστεύω πραγματικά ότι η, δική μας συμβολή θα είναι πολύ σημαντική για την υλοποίηση αυτών των προτεραιοτήτων. Τώρα θα ήθελα να στραφώ στην Ενεργειακή Ένωση και στη συνέχεια και στα ζητήματα ανταγωνιστικότητας. Πρώτον για την ενέργεια. Από τη δική μου σκοπιά η πολιτική ενέργεια είναι πολύ σημαντικό τομέα των κοινών εργασιών και συμφωνιών μα. Συνεχώ και καθημερινά καταναλώνουμε ενέργεια, πολύ συχνά χωρί να το συνειδητοποιούμε. Γι' αυτό η ασφαλή, ε, προσιτή και βιώσιμη ε, αλυσίδα εφοδιασμού είναι κάτι σημαντικό για την ευημερία όλων μα, αλλά και για την ανταγωνιστικότητα τη Ευρωπαϊκή βιομηχανία και την οικονομική ανάπτυξη. Το 2016 έχει οριστεί ω το έτο ε, τη επίτευξης των στόχων από την Ενεργειακή Ένωση και ο στόχο μα είναι πραγματικά να υλοποιήσουμε αυτό το στόχο. Μετά την εξαιρετική δουλειά που πραγματοποίησε η Ολλανδική Προεδρία και με βάση και με το πρόγραμμα εργασιών τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επικεντρωθούμε σε σημαντικές προτάσεις που συνδέονται ε, με τις πέντε βασικές ε, ε, διαστάσεις της Ενεργειακής Ένωσης. Ενίσχυση αρχικά της αλληλεγγύης και της εμπιστοσύνης. Θέλουμε να εξετάσουμε μέτρα που απαιτούνται για την για, προκειμένου οι οικονομίες μας να φύγουν από την οικονομία του άνθρακα σε ένα, με έναν οικονομικά αποδοτικό τρόπο, ενώ παράλληλα θα βελτιώνουμε και την ενεργειακή αποδοτικότητα και ανταγωνιστικότητα θέλουμε ε, να διεξαγάγουμε διαπραγματεύσεις με ένα ανοιχτό και δίκαιο τρόπο και με μια ισορροπημένη προσέγγιση στους τρεις πυλώνες της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής. Οι στόχοι της ΕΕ Ένωσης ε, είναι κάτι που στηρίζεται από το Συμβούλιο ε, συστηματικά και γι' αυτό θέλουμε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνεχίσει να συμβάλλει με πολύ ενεργό τρόπο. Έχουμε πολλούς σημαντικούς φακέλους επιτάπητος και η Ευρωπαϊκή Τροπή ε, έχει ακόμα ορισμένα σχέδια τα οποία θα δημοσιοποιήσει μέσα στην επόμενη χρονιά. Χαιρόμαστε ιδιαίτερως που ο τριμερής διάλογος της 15 ε, Ιουνίου επέτυχε μια πολιτική συμφωνία που έχει ήδη επικυρωθεί ε, στα τέλη Ιουνίου. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και την εισηγήτρια κυρία Κάπελ και τους σκιώδεις και όλους τους ε, συμμετέχοντες ε, σε ένα εξαιρετικό παράδειγμα πολύ αποτελεσματικής ε, διοργανικής συνεργασίας. Τώρα, θα ήθελα επιγραμματικά να συνοψίσω τι προθέσει μα στου επιμέρου φακέλου. Το Συμβούλιο υιοθέτησε τη Γενική Προσέγγιση για την πρόταση αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου για την σήμαση ενεργειακή αποδοτικότητα το 2015 υπό την Προεδρία του Λουξεμβούργου. Χαιρετίζουμε την εντολή που έχει δοθεί ε, στον εισηγητή και θεωρούμε ότι θα μας επιτρέψει να επιτύχουμε μια ταχύτατη ε, συμβαστική λύση με προσθεθμένη αξία και για τους πολίτες και για τη βιομηχανία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε το αποκαλούμενο πακέτο ασφάλειας ε, για το φυσικό αέριο, που περιλαμβάνει δύο νομοθετικέ προτάσεις για την ασφάλεια φωδιασμού αερίου και για ε, συμφωνίε συμφωνίες στον τομέα τη ενέργειας τον Φεβρουάριο τρέχοντος. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν υψηλό επίπεδο φιλοδοξιών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, και χαιρετίζουμε τον διορισμό των δύο εισηγητών γιατί και αυτό το θέμα βρίσκεται ε, στις βασικές μας προτεραιότητες. Σε ό,τι αφορά τι διακυβερνητικέ συμφωνίε δομέα τη ενέργεια, θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και αυξημένη ε, διαφάνεια. Ωστόσο, βλέπουμε ότι και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπάρχουν αποκλίνουσε απόψει ω προ τον τρόπο επίτευξη αυτού του στόχου. Ωστόσο, η Ολλανδική Προεδρία ε, μας οδήγησε σε μια συμβαστική λύση που οδήγησε με τη σειρά της σε μια γενική προσέγγιση στο Συμβούλιο του 2016. Θεωρώ ότι η συμβαστική λύση ε, με βάση την εξάντε αξιολόγηση των ε, διακυβερνητικών συμφωνιών φυσικού αερίου είναι πολύ σημαντική κίνηση και βελτίωση σε σχέση με το εφιστάμενο σύστημα και θα πρέπει έτσι να την βλέπουμε. Ε, η ασφάλεια φωτιασμού ω προ το φυσικό αέριο αποτελεί ακόμα θέμα για πολλέ περιφέρειε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει ο αναφερμένο κανονισμό. Ε, βλέπουμε μάλλον ότι έχει πολλά ανοιχτά και εκκρεμία ακόμα ζητήματα όπου ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί θέση του Συμβουλίου. Αυτό συμπεριλαμβάνει και την λεγγύη και την βριακή συνεργασία καθώ και τη διαφάνεια των ε, συμβάσεων φυσικού αερίου. Προσβλέπουμε σε έναν επικοδομητικό διάλογο με το Κοινοβούλιο για αυτά τα ζητήματα. Σκοπός μας είναι να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσει το συντομότερο δυνατόν. Σε ό,τι αφορά του ε, φακέλους ε, ενεργειακής ε, απόδοσης που θα δημοσιοποιηθούν το φθινόπωρο, σκοπός μας είναι να διοργανώσουμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων με το Συμβούλιο και να γίνει μια συζήτηση πολιτικής στο Συμβούλιο Ενέργειας το Δεκέμβρη σημαντική δέσμη προτάσεων για την διακυβέρνηση της Ενεργικής Ένωση, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τον νέο σχεδιασμό τη αγορά, ε, θα δημοσιοποιηθούν ε, μόλις τα τέλη της δική μας Προεδρίας και έτσι η επόμενη Προεδρία της Μάλτα θα είναι αυτή που θα αναλάβει ε, τις διαπραγματεύσεις αυτούς του φακέλου, που θεωρώ ότι θα είναι εξαιρετικά σημαντική για το μέλλον τη Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική. Όμως, ε, θα προσπαθήσουμε και εμεί να ανοίξουμε τον δρόμο για αυτέ τι ε, συζητήσει, όπω έχει συμφωνηθεί από το πρόγραμμα των, του Τρίτων Προεδριών. Οι Ολλανδοί συνάδελφοι ήδη έκαναν κάποιε συζητήσει για τον ε, σχεδιασμό τη αγορά και εμεί θα συζητήσουμε τα θέματα τη ε, διακυβέρνηση στο, στο άτυπο Συμβούλιο Ενέργεια αύριο στην Βρατισλάβα. Θα εξετάσουμε τι τιμέ και το κόστο τη ενέργεια, καθώ και την ενεργειακή ασφάλεια στο πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το Ευρωπημένο Φυσικό Αέριο και χαίρομαι ιδιαίτερως, κύριε Πρόεδρε, που δεχθήκατε την πρόσκλησή μας να μιλήσετε σε αυτή την διοργάνωση. Η Ενεργειακή Ένωση είναι επίσης θέμα καλύτερης συνεργασίας και μεταξύ περιφερειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και των ε, διεθνών μας εταίρων. Θέλουμε να δούμε πώς θα ενισχύσουμε τη σχέση μας με μεγάλους παρόχους ενέργειας, κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε και την ενεργειακή μας ασφάλεια. Μεγάλη προσοχή θα ευαισθησούμε και ε, στην περιοχή της ε, Ανατολικής, ε, Νότια Ανατολικής Ευρώπης και χώρες της ενεργειακής κοινότητας. Είναι κάτι το οποίο έχει, η σημασία αυτής της περιφέρειας μάλλον έχει τονιστεί και από την πρόσβατη δήλωση Ευρωβουλευτών. Η πυρηνική ενέργεια τώρα διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο ενεργειακό μείγμα πολλών ε, κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό πρέπει να διασφαλίσουμε την χρήση ασφαλού και βιώσιμη ε, ε, χρήση πυρηνική ενέργεια που θα συμβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια και θα αντιμετωπίζει και τα θέματα κλιματική αλλαγή. Ένα από τα πλέον συζητημένα ζητήματα είναι ε, το πρόγραμμα PINK πυρηνικής Ε, και είναι κάτι το οποίο χαιρετίζει η Σλοβακική ε, Προεδρία, την ανακοίνωση δηλαδή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το πρόγραμμα PINK θα συστηθεί και στην επερχόμενη ε, συνδιάσκεψη πυρηνικής ενέργειας στην Πρωτισλάβα στις αρχές Οκτωβρίου. Το δεύτερο θέμα το οποίο θέλω να, στο οποίο θέλω να αναφερθώ σήμερα είναι η ανταγωνιστικότητα. Θεωρούμε ότι η ανταγωνιστικότητα και η καινοτομία είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Θεολογίου για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Είναι απαραίτητο οι εταιρείε να έχουν στην διάθεσή του τι βέλτιστε δυνατέ ε, συνθήκε προκειμένου να λειτουργούν, ιδιαίτερα όταν θέλουν να επιτύχουν στον ε, διεθνή ανταγωνισμό. Η πρόσφατη κρίση στον τομέα του Χάλαβα, Χάλιβα και οι ολοένα και ισχυρότερε φωνέ από άλλε βιομηχανίε και άλλου κλάδου αποδεικνύουν ότι στην Ευρώπη δεν είμαστε πάντοτε ικανοί να παρέχουμε το καλύτερο ρυθμιστικό και επιχειρηματικό περιβάλλον προκειμένου να αναπτύσσεται η βιομηχανία. Πρέπει γι' αυτό λοιπόν να συνδράμουμε και να ε, ενώσουμε τι δυνάμει μα προκειμένου να προστατεύσουμε την ευρωπαϊκή βιομηχανία στην Ευρώπη. Θεωρούμε ότι η βιομηχανία ε, είναι ένα πολύ κρίσιμο τομέα στι οικονομίε μα. Επίση πιστεύουμε ότι θα πρέπει ως Προεδρία να προωθήσουμε το στόχο που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το 20% του ΑΕΠ στην Ευρώπη να προέρχεται από τη βιομηχανία. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, θα επικεντρωθούμε σε τρεις συγκεκριμένους τομείς. Πρώτον, εξυγχρονισμός της ευρωπαϊκής βιομηχανίας η ψηφιακή μεταμόρφωση και ο μετασχηματισμός αυτός της βιομηχανίας, ιδιαίτερα στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ε, έχει καθυστερήσει σε σύγκριση με τους παγκόσμιους ανταγωνιστές μας. Προτεραιότητά μας είναι λοιπόν να υποστηρίξουμε την εφαρμογή ε, και την υλοποίηση αποτελεσματικών μέτρων στον τομέα αυτό. Θα επικεντρωθούμε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον, ε, όσον αφορά την, ε, τον συντονισμό εθνικών και περιφερειακών πρωτοβουλειών για την ψηφιοποίηση των βιομηχανιών μας. Πιστεύουμε ότι η προσπάθεια αυτή μπορεί να επιφέρει πολλές συνέργειες και να διευκολύνει τη διαδικασία εξυγχρονισμού της βιομηχανίας. Προκειμένου να υποστηριχθεί η διαδικασία αυτή, πρέπει επίση να εξασφαλίσουμε ότι το εργατικό δυναμικό θα έχει τα κατάλληλα προσόντα και τι κατάλληλε δεξιότητε. Φιλοδοξία μα είναι να αντιμετωπίσουμε το έλλειμμα ψηφιακών δεξιοτήτων σε ολόκληρη την Ευρώπη, ενθαρρύνοντα την βιομηχανία να συνεργαστεί με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, προκειμένου όλοι μαζί να καταστούν πρωτοπόροι σε αυτήν την πρωτοβουλία για τι δεξιότητε. Επιπλέον, θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα του εξοχρονισμού τη βιομηχανία Κατά την ε, άτυπη συνδιάσκεψη των ε, Υπουργών που είναι αρμόδιοι για την ανταγωνιστικότητα που θα γίνει την επόμενη ε, εβδομάδα στην Πρατισλάβα. Ο δεύτερος τομέας μας είναι το να τεθεί στο επίκεντρο η ανταγωνιστικότητα. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις ε, στον τομέα της ανταγωνιστικότητας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ε, και με την έγκριση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προτείνει να τεθεί η ανταγωνιστικότητα ω μια κεντρική διάσταση σε, όλες τις, σε όλους πολιτικής και μάλιστα πολύ πολύ ψηλά πάνω στην ατζέντα. Αυτό σημαίνει ότι κάθε πολιτική και κάθε σχετική πρόταση θα πρέπει να μην εμποδίζει την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των επιχειρήσεών της και αυτή η διάσταση θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Θέλουμε να συνεχίσουμε τι προσπάθειε που έχουν ήδη γίνει από τι προηγούμενε προεδρίε. Η Σλοβακική Προεδρία φιλοδοξεί να βασιστεί σε, στον τομέα αυτό προκειμένου να ωφεληθούν όλες οι ευρωπαϊκές εταιρείες. Σκοπός μας είναι να προτείνουμε πολιτικές σε αυτούς τους, τομέα, τομείς ε, που είναι πολύ σημαντική για την ανταγωνιστικότητα και συγκεκριμένα πέραν από την Ενεργειακή Ένωση που σας ανέφερα ήδη, μιλώ για την ψηφιακή, για την ενιαία αγορά, με συγχωρείτε, για την ψηφιακή ενιαία αγορά και το θεματολόγιο για την καλύτερη νομοθεσία. Επιπλέον, θέλουμε να κάνουμε και κλαδικούς τομεακούς ε, διαλόγους στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και ταυτόχρονα θα ήθελα ε, να, να, αναφερθώ στον ε, τομέα του Χάλιβα που όπως είπα, όπως είπα και νωρίτερα αντιμετωπίζει μεγάλες ε, προκλήσεις αλλά και στον τομέα της εμπορικής πολιτικής ή στην πολιτική για την κλιματική αλλαγή έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε. Διαδικασίες αντι-dumping, μελλοντική απόφαση για το MES China, EU ATS κτλ. Και τέλος, ε, σας έχω αναφέρει ήδη τον ε, τομέα του Χάλβα, αλλά θα ε, επικεντρωθούμε, θα δώσουμε τη δέουσα προσοχή και στις ενεργοβόρες βιομηχανίες. Στο, το θέμα αυτό μάλιστα θα συζητηθεί και στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας, ε, όπως είπα και την επόμενη εβδομάδα. Θα γίνει στην Πρατισλάβα να σας δώσω λίγες περισσότερες πληροφορίες για το τι έχουμε εμεί κατά νου στους άλλους τομείς ε, κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας, συγκεκριμένα ε, και που σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και καλύτερη νομοθεσία. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα ήθελα να τονίσω ότι προκειμένου να ε, στεφτεί με επιτυχία το θεματολόγιο για την ανταγωνιστικότητα θα πρέπει να ληφθούν σοβαρότατα υπόψη οι επιπτώσεις του στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το να προωθηθεί λοιπόν ένα καλύτερο νομοθετικό πλαίσιο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι αναπόσπαστο στοιχείο των δικών μας προτεραιοτήτων, της Προεδρίας της Σλοβακίας. Στο πλαίσιο λοιπόν του, του, του, του ισχύοντος ε, πλαισίου πολιτικής, ε, εμείς ε, και στο, τομέα, και στο πλαίσιο μάλλον της ενιαίας αγοράς αλλά και της ψηφιακής ενιαίας αγοράς θεωρούμε ότι έχει σημασία να προωθηθούν διάφορε πρωτοβουλίε προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επίση, Χρειάζεται να διευκολύνουμε την πρόσβαση αυτών των επιχειρήσεων στι αγορέ, να καταστήσουμε και να δημιουργήσουμε, να θεσπίσουμε ένα καλύτερο νομοθετικό πλαίσιο και να προωθήσουμε τι δεξιότητε. Θα γίνει και μια σχετική σύνοδο μικρομεσαίων επιχειρήσεων τον Νοέμβριο στην Πραστιτσλάβα, όπου θα συζητηθούν όλα αυτά τα θέματα σε βάθο. Όσον αφορά την καλύτερη νομοθεσία και το σχετικό θεματολόγιο, το, την, την καλύτερη και τη μελλοντοστραφή νομοθεσία, δηλαδή η οποία θα επιτρέπει την κοινοτομία, αυτό το θέμα αποτελεί μια απόλυτη προτεραιότητα για τη Σλοβακία γιατί είναι απαραίτητο προκειμένου να δημιουργηθεί η επιδιωκόμενη οικονομική ανάπτυξη και η ενίσχυση της απασχόλησης. Χρειάζεται λοιπόν να εξετάζουμε σοβαρά το ζήτημα της ποιότητας των νομοθετημάτων που θεσπίζουμε και όχι να ε, επιφορτίζουμε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μας με περιττό βάρος. Θα συνεχίσουμε λοιπόν τις, προτε... τις προσπάθειές μας ε, σε αυτόν τον τομέα και ε, σε αυτό το τομέα θα ήθελα να αναφερθώ και στα εκρεμή ζητήματα όσον αφορά τη διοργανική συμφωνία για την ε, καλύτερη νομοθεσία. Κύριε Πρόεδρε, ε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής ε, και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Σλοβακική Προεδρία και οι συνάδελφοί μου είμαστε έτοιμοι να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια προκειμένου να ε, δημιουργήσουμε και να αναπτύξουμε και να επιτύχουμε θετικά και απτά αποτελέσματα στον τομέα της ενεργειακής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ανταγωνιστικότητα εμείς θα ε, προσέλθουμε στις διαπραγματεύσεις λοιπόν με ειλικρίνεια και με επικοδομητικό πνεύμα. Θα σας, ευχαριστούμε, ε, σας ευχαριστώ που θα μοιραστείτε μαζί μου τις δικές σας απόψεις και θα μου πείτε τις δικές σας γνώμες σχετικά με το πρόγραμμα της Σλοβακικής Προεδρίας που μόλις σας παρουσίασα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Εμείς σας ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας. Βεβαίως είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με την Σλοβακική Προεδρία και ευχαριστούμε και ε, για την ε, ε, γενικότερα θετική σας στάση γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που σας βλέπουμε και εγώ και οι συνάδελφοί μου και μάλιστα και διάφοροι πρόεδροι επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκτιμούν ιδιαίτερο τη στάση της Σλοβακικής Προεδρίας. Θα δώσω τώρα το λόγο στους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες, η κυρία Βέρνερ. Ευχαριστώ. Κιόλας, ε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ για την παρουσίασή σας και για την ετοιμότητά σας να συνεργαστείτε μαζί μας στενά. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό σε αυτές τις ε, εποχές που ζούμε και να έχουμε όλοι μαζί την δυνατότητα να προσφέρουμε στους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης και πραγματικές λύσεις. Και με αυτό έρχομαι στο πρώτο θέμα που με ενδιαφέρει, στον τομέα της ενεργειακής πολιτικής. Ε, όπως είπατε, ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του τριμερούς διαλόγου όσον αφορά την ενεργειακή επισήμιση και η δική μας ε, άποψη πολιτική ομάδα, όπως δηλώσαμε και εδώ στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια, είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει γρήγορα ένα descaling, προκειμένου το ταχύτερο δυνατό να οι καταναλωτές να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό το νέο σήμα, σε αυτή τη νέα σήμανση από το α έως το G και από ό,τι άκουσα οι απόψεις ε, στο Συμβούλιο είναι πολύ πιο ήπιες, θεωρούν στο Συμβούλιο ότι θα πρέπει να διαρκέσει η διαδικασία πολύ περισσότερα χρόνια από ό,τι θα θέλαμε εμείς τουλάχιστον. επομένω θα ήθελα να μου πείτε εσείς ποια είναι η δική σας γνώμη, πώς βλέπετε να, να εξελίσσονται αυτές οι διαπραγματεύσεις και πόσο έτοιμοι είστε να μπείτε σε συμβιβασμού. Επίση, ε, καλό είναι το ότι αναφερθήκατε στο στόχο του 20%. Πρόκειται για ένα στόχο της απερχόμενης, της απελθούσας μάλλον κομισιόν. Νομίζω όμως ότι είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα αυτό το να τεθεί αυτός ο στόχος του 20% ΑΕΠ στην Ευρώπη από τη βιομηχανία και πρέπει να, να, να δοθεί σε αυτό το στόχο ε, ιδέως προτεραιότητα. Παρόλα αυτά όμως νομίζω ότι δεν πρέπει να ακολουθήσουμε μια οριζόντια προσέγγιση για όλη την οικονομία αλλά αντίθετα να εξετάσουμε ανακλάδο τις επιχειρήσεις για να καθορίσουμε και τις ανάγκες των επιμέρους κλάδων και των επιμέρων, επιμέρους ε, ε, επιχειρήσεων. Άρα η δική σας γνώμη, κατά πόσο πιστεύετε ότι είναι εφικτή μια τέτοια προσέγγιση, κάθετη και όχι οριζόντια. Ε, μάλιστα πρόσφατα εδώ στο Κοινοβούλιο ε, ψηφίσαμε και ένα, ε, εγκρίναμε και ένα ψήφισμα για τους σιδηροδρόμους. Θα θέλαμε λοιπόν τη δική σας γνώμη. Τρίτον, όσον αφορά το καθεστώς αγοράς της Κίνας και την, τον χειρισμό αυτού του θέματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και την συμφωνία με τις, ε, ε με τις ΕΙΠΑ, ε, ε, μάλιστα υπάρχει, με υπάρχει ε, πρόσφατα μια δήλωση εν, εν, μιας μεγάλης χαλιβουργίας της Σλοβακίας για το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αναλάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα αντι-dumping προκειμένου να προστατευτεί η χαλιβουργία της Ευρώπης ε, από το dumping που δέχεται από την Κίνα. Ποιες είναι λοιπόν οι ιδέες οι δικές σας και οι γνώμες σας σχετικά με αυτό το θέμα. Εκ μέρους του ΕΛΚ λέει ο Πρόεδρος, κυρία Ζαμπόρσκα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ. Και εγώ ε, προέρχομαι από την ε, Σλοβακία και επομένως ε, είμαι πολύ ευτυχής που σας υποδεχόμαστε εδώ στην Επιτροπή Ήτρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω γιατί αναφερθήκατε στο πρόγραμμα της Σλοβακικής Προεδρίας. Τα ζητήματα τα οποία αναφέρατε είναι ιδιαίτερως επίκαιρα και μας απασχολούν και εδώ στην Επιτροπή μας ιδιαίτερος. Δύο ερωτήσεις να σας υποβάλω κύριε Υπουργέ. Είμαι... Είμαι και εγώ σκιώδης ε, εισηγήτρια για το θέμα της αγοράς ε, και θέλω να ρωτήσω ε, ποια είναι για την κυκλική οικονομία συγγνώμη, και ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η θέση της Λογικής Προεδρίας όσον αφορά το ζήτημα αυτό της ε, κυκλικής οικονομίας. Δεύτερο, γίνεται αναφορά στην ε, εμβάθυνση της ε, νομισματικής ε, ένωσης και της ενιαίας αγοράς και όσον αφορά και όσον αφορά και την νομισματική ένωση και την δημοσιονομική ένωση. Θέλετε να μας πείτε τι σκοπεύει να κάνει η Σλοβακική Προεδρία όσον αφορά τη μεγαλύτερη διασύνδεση των προϋπολογισμών. Όσον αφορά Εξ ονόματος ε, των συντηρητικών, παρακαλώ κύριε συνάδελφε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω και εγώ σλοβακικά. Συμφωνώ λοιπόν με τον ε, συνάδελφο ότι είναι μεγάλη μας τιμή που λίγες μέρες αφού το ανέλαβε η χώρα μας στην Προεδρία βρίσκεστε εδώ. Η Επιτροπή μας λοιπόν εδώ είναι μια πολύ σημαντική Επιτροπή γιατί μιλούμε για την βιομηχανία και την ενέργεια σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με μεγάλο λοιπόν ενδιαφέρον παρακολούθησα την παρουσίαση του προγράμματος της Σλοβακικής Προεδρίας και αυτά που είπατε κύριε Υπουργέ, Υπουργέ θεωρώ ότι χαρακτηρίζονται από έναν πραγματισμό και έναν ρεαλισμό και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γνωρίζουμε όλοι πόσο περίπλοκες είναι οι εποχές στις οποίες ζούμε, όχι μόνο λόγω του Brexit, για την Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή, αλλά και λόγω των ε, σχέσεων ε, με τις ΗΠΑ, αλλά και όσον αφορά το καθεστώς οικονομίας της αγοράς της Κίνας. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σύνθετα και περίπλοκα θέματα και είμαι πολύ χαρούμενος που αναφερθήκατε και στο ζήτημα της Ενεργειακής Ένωσης όσον αφορά την ε, ασφάλεια εφοδιασμού ε, ενέργειας. Το πρώτο μου ερώτημα λοιπόν είναι το εξής. Ακριβώς επειδή από την εμπειρία της Σλοβακίας ε, γνωρίζουμε ότι έχετε μεγάλη πείρα σε αυτό τον τομέα, είστε χώρα διέλευσης και έχετε, ε, βρίσκεστε πολύ κοντά, βρισκόμαστε πολύ κοντά ως χώρα στην Ουκρανία και στην Ρωσία. Πώς μπορούμε λοιπόν να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες για τη διάθεση του LNG στην αγορά, ε, ποια θα είναι τα εμπόδια και τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, ε, χαίρομαι πολύ που ε, θεωρείτε ότι το θέμα αυτό έχει πολύ ψηλή προτεραιότητα. Επίσης, αυτό που, αναφερθήκατε, αυτό που αναφέρατε όσον αφορά τον εξυγχρονισμό της ευρωπαϊκής βιομηχανίας είναι και αυτό ένα πάρα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Ε, έχουμε μπροστά μας μια πολύ ε, ευρεία διαδικασία εξυγχρονισμού και ψηφιοποίησης. Ε, ποια λοιπόν πιστεύετε ότι θα είναι η κατάσταση, ποιο θα είναι λοιπόν μάλλον το καθεστώς το οποίο θα αποδοθεί στην Κίνα. Ακριβώς διότι το θέμα αυτό θα συζητηθεί ιδίως προ το τέλος της Συλλοβακικής Προεδρίας και γνωρίζουμε όλοι το θέμα αυτό, είναι κάθε άλλο παρά Άρα μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να μάθουμε ε, ποια θα είναι η στάση της δικής σας χώρας ε, στο θέμα αυτό. Είναι πάρα πολύ περίπλοκο το θέμα, δεν μπορούμε να το προσεγγίσουμε με όρους άσπρο ή μαύρο και θα έχουμε πολύ έντονες συζητήσεις. Και νομίζω ότι όλα αυτά θα καταλήξουν σε κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα στο τέλος του χρόνου, όπως είπα, οπότε αξίζει να το συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ λοιπόν κύριε Υπουργέ για όλα όσα είπατε. Γνωρίζουμε ότι είναι πολύ σημαντικές οι εμπειρίες που έχει συλλέξει η Σλοβακία. Και ότι σε αυτήν ακριβώς την εμπειρία της Σλοβακίας μπορούμε να βασιστούμε για να χαράξουμε και τι μολυντικέ μα πολιτικέ. Θα ήθελα εκ μέρους ολόκληρης πολιτική μα ομάδα να σα ευχηθώ κάθε επιτυχία στο έργο σα, γιατί γνωρίζω ότι και έξι μήνες είναι χρονικό διάστημα πολύ μικρό. Αν δεν συνυπολογίσει κανείς ότι σε αυτό θα χάσουμε και τους δύο μήνες του καλοκαιριού, έχετε πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή σας, αλλά από τη δική μας πλευρά μπορώ από, από τη θέση μας σας διαβεβαιώσω ότι θα έχετε κάθε υποστήριξη από εμάς η κυρία Κάλλας, εξ ονόματος της Άλντε, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίασή σας. Είπατε ότι έχετε δύο προτεραιότητες ως Σλοβακική Προεδρία. Ε, το ένα είναι η ψηφιακή αγορά και το άλλο η ενέργεια. Ε, κατά την άποψή μου υπάρχει διασύνδεση ανάμεσα στα δύο θέματα. Όταν μιλάμε για την ψηφιακή ένωση, ε, οπωσδήποτε υπονοούμε ότι χρησιμοποιούμε ή πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα ψηφιακά εργαλεία και στον τομέα της ενέργειας. Ποιες είναι λοιπόν οι απόψεις όσον αφορά το θέμα αυτό. Μια δεύτερη ερώτηση τώρα, η οποία σχετίζεται με αυτά που αναφέρατε για την ενέργεια. Είπατε ότι θέλετε να εστιάσετε την προσοχή σας ε, ε, στην τιμολόγηση της ενέργειας. Τι σημαίνει όμως αυτό. Σημαίνει ότι θα μας υποβάλλετε κάποιο κανονισμό για τη δημολογική πολιτική ή κάτι άλλο. Ε, ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Ρόμπελ Μπερνέρο, εξ ονόματος της ΓΚΟΕ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την παρουσία σας. Εγώ θα επικεντρώσω την παρουσίασή μας σε δύο, στην παρουσίασή μου σε δύο βασικά θέματα, τη βιομηχανία και την ενέργεια. Ε, αναφέρομαι στις ε, συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου και το σχέδιο Juncker. Ε, διαρροές όσον αφορά το TTIP και όσον αφορά το τελικό κείμενο της συμφωνίας ε, ΣΕΤΑ ε, επιβεβαιώνει τους φόβους μας ότι δηλαδή η Κομισιόν θέλει να ε, χρησιμοποιήσει αυτές τις συμφωνίες έτσι ώστε να προωθήσει ε, την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο που παράγονται μέσω της μεθόδου της υδρορογμάτωσης. Ε, δηλαδή θέλει να στηρίξει και να προωθήσει στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των, των, της διατησίας και των διαδικασιών διατησίας στις οποίες θα προσφύγουν οι πολυεθνικές εταιρείες αυτές τις πρακτικές τις οποίες μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήθελε. Ε, στις ε, δικές σας ε, προτεραιότητες πολύ λίγα πράγματα είδα όσον αφορά την, την, εμπορική, την ενεργειακή απόδοση. Τίποτα δεν είδα όσον αφορά τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας. Ερωτώ λοιπόν εσείς ε, θα στηρίξετε την άποψη ότι σε κάθε χώρα μέλος ε, θα υπάρχει η δυνατότητα να μπλοκαριστούν αυτού του είδους οι συμφωνίες μέχρι ότου να έχει ακουστεί η φωνή των Ευρωπαίων πολιτών εάν και εφόσον δεν συμφωνούν με αυτές τις συμφωνίες. Δεύτερον, ε, ποια θα είναι η στάση σας όσον αφορά την μείωση των, της χρήσης και της εισαγωγής των ορυκτών μορφών ενέργειας ε, οι οποίοι, που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάνοντας κοινωνικό και άλλο dumping. Δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε ε, την απελευθέρωση της, ε, του εμπορίου με την Κίνα. Γιατί στην ουσία αυτή η διαδικασία θα οδηγήσει σε ντάμπινγκ κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό. Δεύτερον, το σχέδιο Juncker πέρα από τις, ε, ε, τη μεγάλη ικανοποίηση που πολλοί εξέφρασαν ε, θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα προβλήματα τα οποία εισάγονται μέσω αυτού του προγράμματος στην ουσία κοινωνικοποιούνται οι ιδιωτικοί κίνδυνοι στην ουσία δηλαδή δίνουμε την δυνατότητα στις μεγάλες εταιρείες, στις ιδιωτικές εταιρείες να διαβρώσουν τον κοινωνικό ιστό. Ρωτώ λοιπόν πώς είναι δυνατότητα δυνατόν ευρωπαϊκοί πόροι να χρησιμοποιούνται έτσι ώστε ε, να ε, χρησιμοποιούνται τα χρήματα αυτά τα ευρωπαϊκά ε, για τους κερδοσκόπους και για τη διάσωση τραπεζών και όχι να προωθούνται για κοινωνικούς λόγους και για, την Ευρωπα... για τους πολίτες της Ευρώπης. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ταμπουράνο. Σας χαιρετώ κύριε Υπουργέ. Και εγώ θα ήθελα να υποβάλω τις ερωτήσεις που πρόλαβαν να υποβάλουν ε, οι συνάδελφοι όσον αφορά ε, το TTIP ε, σε σχέση και με το Brexit και με την ενδεχόμενη συμφωνία για το καθεστώς ελεύθερης αγοράς στην Κίνα. Ε, και φυσικά και την εισαγωγή ενεργειακών προϊόντων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, που έχουν παραχθεί με τρόπους απολύτως αντίθετους ε, με τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι οι συμφωνίες ελεύθερης ε, αγοράς και ελεύθερου εμπορίου είναι κάτι που μας απασχολεί όλους ε, και είδαμε και διαρροές ε, του, από το TTIP που εάν επιβεβαιωθούν ε, θα πρέπει να μας πείτε ποια είναι η άποψή σας ε, γιατί εδώ μιλάμε για σύγκληση ενεργειακή ε, η οποία αντιτίθεται πλήρως στις αρχές Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, εδώ επίσης ε, μιλάμε για μια θεσμική διαδικασία η οποία αφορά τις 28 χώρες μέλη και εμπλέκει και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ε, και την Κομισιόν που φαίνεται ότι έχουν πρόβλημα να βρουν ένα κοινό ε, ε, κείμενο. Απ' την άλλη πλευρά ε, μια ενεργειακή επισήμανση η οποία θα είναι μια ετικέτα η οποία θα είναι ίδια για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό σημαίνει μια συγκεκριμένη διαδικασία αφενός ευρωπαϊκή αλλά και συμπερίληψη της άποψης της δικιάς μας ημών των Ευρωβουλευτών που εκπροσωπούμε βεβαίως τους πολίτες της Ευρώπης. Εάν λοιπόν αυτή η διαρροή επιβεβαιωθεί. Θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η θέση σας όσον αφορά το θέμα αυτό. Uh, Σας ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε. is, uh, Κύριε Υπουργέ, ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος των ερωτήσεων. Παρακαλώ αν θέλετε να απαντήσετε. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Για το πρώτο ερώτημα, να απαντήσω στην κυρία Βέρνερ. Σας ευχαριστώ πολύ για το ερώτημά σας. Ε, θα προσπαθήσω να απαντήσω στη μητρική μου γλώσσα όλες τις ε, ερωτήσεις, αλλά στη συνέχεια. Σε εσάς θα απαντήσω στα γερμανικά. Ρωτήσατε λοιπόν ε, για την επισήμανση. Για το δεύτερο ερώτημα, αφορούσε ε, το ποσοστό, το 20% δηλαδή της βιομηχανίας στην οικονομία και το τρίτο αφορούσε το καθεστώς ε, ε, ελεύθερης αγοράς για την Κίνα. Επιτρέψτε μου για το θέμα της επισήμανσης να πω τα εξής. Η πρόταση κανονισμού είναι κάτι το οποίο εμείς εξετάζουμε και θεωρούμε ως θετικό στοιχείο προς την απλούστευση της σύγκρισης ε, της ενεργικής απόδοσης επιμέρους ε, συσκευών από τους πολίτες. Ο σκοπός μας και η φιλοδοξία μας είναι η διαπραγμάτευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, για να γίνουν όλα αυτά με επικοδηματικό τρόπο και να υπάρξει πολιτική συμφωνία το μέτρο δυνατόν. Ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι θα γίνει αυτό και ότι θα είμαστε σε θέση ε, να οικοδομήσουμε σχέσεις ευρύτερης εμπιστοσύνης ε, μεταξύ ε, του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου εν ώψη και άλλων προτάσεων που συνδέονται με την Ενεργειακή Ένωση. Η γενική προσέγγιση που υιοθετήθηκε στις 26 Νοεμβρίου του περασμένου έτους από το Συμβούλιο αποτελεί μια πολύ καλή βάση για περαιτέρω συζητήσει στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας των τριμερών διαλόγων. Εκτιμούμε το έργο που διεκπεραιώνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με επικεφαλή τον κύριο Ταμπουράνο, τον εισηγητή, και χαιρετίζουμε την ε, υιοθέτηση της έκθεσης. Η πρόοδος, οποιαδήποτε πρόοδος μάλλον βασίζεται σε αμοιβαία συνένεση και συμβασμούς και έτσι η Σλοβακική Προεδρία του Συμβουλίου θα προσπαθήσει να εκπληρώσει αυτό το καθήκον με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έχοντας κατά νου όλες τις πιθανές επιπτώσεις και πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε να επιτύχουμε μια συμφωνία που θα είναι αποτελεσματική και θα λαμβάνει υπόψη και τη συνέπειση για τη βιομηχανία. Αυτά για την επισήμανση. Σε ό,τι αφορά το μερίδιο, το 20% τη βιομηχανία ε, επί του ΑΕΠ, ξέρετε, Είμαστε από τις χώρες που έχουν ε, τους μεγαλύτερους αυτούς συντενελεστές, δηλαδή το μερίδιο της βιομηχανίας ε, στο ΑΕΠ, 20%. Και θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό και για το Συμβούλιο και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αυξήσει αυτό το μερίδιο της βιομηχανίας ε, επί του ΑΕΠ και ότι αυτό είναι μια θετική τάση γιατί ιδίως σε τέτοιες εποχές όπως η σημερινή η βιομηχανία ε, μας οδηγεί και συμβάλλει προς ε, την ε, οικονομική βιωσιμότητα αλλά και την ανάπτυξη. Και εμείς από πλευράς μας λοιπόν θα προσπαθήσουμε να στηρίξουμε οποιαδήποτε πρόταση, είτε αυτή προέλθει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα στηρίξουμε λοιπόν οποιαδήποτε τέτοια πρόταση έχει ως στόχο την αύξηση του μεριδίου της μηχανίας στην οικονομία. Σε ό,τι αφορά το καθεστώς ε, ελεύθερης αγοράς για την Κίνα, θεωρώ ότι αυτό το θέμα έχει τεθεί από πολλούς ε, ομιλητές. Νομίζω ότι ο κύριος Τωσενόφσκι, αν δεν κάνω λάθος, ε, το έθιξε προηγουμένως. Και η κυρία Μπερμέχο το έθιξε, καθώς και ο κύριος Ταμπουράνο. Για αυτό το θέμα, πιο συγκεκριμένα, για τη χορήγηση του καθεστώτος ελεύθερης αγοράς στην Κίνα, θα το εξετάσουμε με πολύ μεγάλη προσοχή. Και με τη δέουσα επιμέλεια, λοιπόν, γιατί είμαστε από τις χώρες που σε περίπτωση χορήγηση τέτοιου καθεστώτος ε, στην Κίνα θα ήμασταν ε, ενδεχομένως σε κίνδυνο. Η χώρα μας δηλαδή. Αυτό είναι κάτι το οποίο ε, θα εξετάσουμε σε διάφορα βήματα κατά τη διάρκεια της Λοβική Προεδρίας και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Οκτώβριο και στο Συμβούλιο Υπουργών Εμπορίου τον Νοέμβριο. Και γνωρίζουμε ότι οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να υλοποιηθούν το Δεκέμβριο. Θα έχουμε ιδιαίτερα ενεργό ρόλο στην όλη διαδικασία και οποιαδήποτε λύση κι αν υιοθετηθεί από το Συμβούλιο θα εμεριμνήσουμε για την ε, δέουσα προστασία του ευρωπαϊκού εμπορίου. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα εξεταστεί σε ύψιστο επίπεδο, δηλαδή σε επίπεδο επικεφαλής ε, και αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Και εξ όσων γνωρίζω, η συζήτηση και οι αποφάσεις σχετικά με την χορήγηση αυτού του οικονομικού καθεστώτος ε, στην Κίνα θα πρέπει να υιοθετηθεί ακριβώς ε, σε ύψιστο επίπεδο τον Οκτώβριο κάποια στιγμή. Όπως είπα λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να υιοθετήσουμε τέτοια μέτρα που ε, να μεριμνούν για την επαρκή προστασία της βιομηχανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, κυρία Ζαμπορσκά, σα ευχαριστώ για τι ερωτήσει σα. Σε ό,τι αφορά την κυκλική οικονομία, ίσως δεν είμαι πλέον κατάλληλο ω Υπουργό Οικονομία να απαντήσω σε κάτι τέτοιο. Μάλλον θα πρέπει να απευθύνεται το ερώτημα στον Υπουργό Περιβάλλοντο. Αλλά επειδή και στο παρελθόν έχω διατελέσει Υπουργό Περιβάλλοντο, θα προσπαθήσω να απαντήσω. Θεωρούμε ότι όλα τα μέτρα και οι δέσμε ε, μέτρων για την κυκλική οικονομία θα βοηθήσουν του τομεί και του κλάδου οικονομία που προσπαθούν κάπως να κρατήσουν τη θέση τους στην παγκόσμια οικονομία. Ελπίζουμε ότι και η αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Συστήματος ETS ε θα συμβάλλει όσο επιθυμούμε προς αυτούς τους ε, στόχους για την κλιματική αλλαγή. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα απασχολήσει ε, και στο Συμβούλιο στην Μπρατισλάβα Θα εξετάσουμε λοιπόν τις τιμές της ενέργειας αλλά και την κυκλική οικονομία. Θα μας απασχολήσουν λοιπόν οι κατά την διάρκεια της Προεδρίας μας αυτά τα ζητήματα. Μετά το δεύτερο ερώτημά σας αφορούσε την διασύνδεση ε, επιμέρους ζητημάτων ε, δημοσιονομικών με άλλα. Δεν μπορώ να απαντήσω ε, σε αυτά τα ζητήματα γιατί αφορούν περισσότερο τον Υπουργό Οικονομικών παρά εμένα. Μπορώ να το προωθήσω λοιπόν στον Υπουργό Οικονομικών ή στους συναδέλφους που εργάζονται εδώ στην μόνιμη αντιπροσωπεία και προκειμένου να σας δώσουν μια απάντηση γραπτός. Ωραία. Τώρα θα προσπαθήσω να απαντήσω στα ερωτήματα του κ. Τωσινόφσκη. Σας ευχαριστώ πολύ και για την στήριξη ε, που εκφράσετε προς το πρόσωπό μου. Με ρωτήσατε για το φυσικό αέριο και την διασύνδεση των διαδρόμων φυσικού αερίου. Θέσατε και κάποια ζητήματα σχετικά με το υγροποιημένο φυσικό αέριο, LNG. Θα ήθελα να πω ότι η αλληλεγγύη, ιδίω σε περίοδους κρίσης, θεωρούμε ότι είναι μία από τις ε, βασικότερες αρχές που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν στην κάλυψη ελλείψεων ή και διακοπών σε ό,τι αφορά την αλυσίδα και στην χώρα σας ε, αλλά και στη δική μου, πριν από μερικά χρόνια, για πρώτη φορά σε 40 χρόνια είχαμε διακοπή ε, στο δίκτυο και ήμασταν από τις πρώτες χώρες που έπρεπε να αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα. Και τότε ήταν κέρια σημασία ε, η αλληλεγγύη. Και για πρώτη φορά είχαμε την αντίστροφη ε, ροή φυσικού αερίου, που ήταν κάτι άνευ προηγουμένου τα τελευταία 40 χρόνια. Δεν είχε ε, υλοποιηθεί ποτέ ένα τέτοιο μέτρο μέχρι σήμερα. Βεβαίως, η αλληλεγγύη αυτή και αυτός ο μηχανισμός λαμβάνει υπόψη και τις ιδιαιτερότητες επιμέρους αγορών και εξετάζει και το ζήτημα των αποζημιώσεων. Λίγο πριν τη σημερινή συνεδρίαση μαζί με τον κύριο Μπούζεκ. Συζητήσαμε αυτά τα θέματα του θεματολογίου της, ε, των εφοδιασμού με φυσικό αέριο και εξετάσαμε και αυτό το θέμα της αλληλεγγύης. Ως προς την περιφερειακή συνεργασία, τα κράτη-μέλη έχουν εκφραστεί υπέρ μιας διευρυμένης ευελιξίας σε ό,τι αφορά τη, τον καθορισμό των περιφερειών και σε ό,τι αφορά την υλοποίηση των εθνικών ε, σχεδίων δράσης και των ε, σχεδίων έκτακτης ε, παρέμβασης. Πρέπει λοιπόν να τα εξετάσουμε όλα αυτά από κοινού, γι' αυτό πρέπει να βρούμε μια συμβαστική λύση και αυτό θα είναι καθοριστική εξέλιξη. Ελπίζουμε να προχωρήσουμε όσο γίνεται περισσότερο, να καταλήξουμε δηλαδή σε συμφωνία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και ή δυνατόν να ολοκληρωθεί αυτό το ζήτημα κατά τη διάρκεια τη Προεδρία μα. Σε ό,τι αφορά την περιφερειακή συνεργασία, να σα δώσω ένα παράδειγμα ω προ την κατανομή των χωρών. Η Σλοβακία ήταν στην ίδια κατηγορία με τη Γερμανία, την Τσεχία, την Πολωνία. Βεβαίως αυτή είναι μια καλή συνεργασία βάσει πολλών χρόνων εμπειρία και εφόσον περάσαμε μαζί πολλέ κρίσει. Όμω ορίσαμε ότι πρέπει να συμπεριλάβουμε και χώρε όπω η Αυστρία, Αυστρία ε, σε αυτή τη συνεργασία, γιατί έχουμε πόλει που είναι πολύ κοντά στα σύνορα με τη Σλοβακία. Έτσι θα υπάρχει ακόμα καλύτερη διασύνδεση. Μετά είναι το ζήτημα τη Ουγγαρία, που είναι και γειτονική χώρα αφενό, αλλά και συμμετέχει ε, σε δίκτυα φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Καλό θα ήταν λοιπόν να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία σε ό,τι αφορά το καθορισμό των περιφερειών. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι η φιλοδοξία μας είναι όσο γίνεται να προχωρήσουμε σε αυτές τις διαπραγματεύσεις προκειμένου να ολοκληρωθούν κατά τη διάρκεια της Σλοβακικής Προεδρίας. Για το καθεστώς της Κίνας ήδη απάντησα προηγουμένως. Να απαντήσω στην κυρία Κάλλας. Με ρωτήσατε για την Ενεργειακή Ένωση. και η διασύνδεση μεταξύ ενέργειας και ψηφιακής οικονομίας. Αλλά με ρωτήσατε και για τις ε, τιμές, για το κόστος της ενέργειας θεωρούμε την Ενεργειακή Ένωση μία ευκαιρία για την διαμόρφωση συνεργειών μεταξύ επιμέρου τομέων. Κλιματική πολιτική, ενεργειακή πολιτική, ψηφιακή πολιτική και ψηφιοποίηση. Η επίτευξη αυτών των ε, στόχων θα πρέπει να συνοδεύεται και από μια οικονομική απόδοση, λαμβάνοντας υπόψη και την ανταγωνιστικότητα και σε ό,τι αφορά τις τιμές της ενέργειας. Αύριο και μεθαύριο, όπως προανέφερα, θα έχουμε άτυπη ε, υπουργική διάσκεψη στην Πρατισλάβα. Και ένα από τα θέματα θα είναι ακριβώς οι τιμές ε, της ενέργειας και η προσβασιμότητα επίσης. Θα μας απασχολήσουν λοιπόν ε, ιδιαίτερως αυτά τα ζητήματα κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας. αλλά και για τα περιβαλλοντικά και κλιματικά ζητήματα. Θα προσπαθήσουμε να διαμορφώσουμε τις προϋποθέσεις, ούτω ώστε σταδιακά η κοινωνία μας ε, να κινηθεί προς ε, μια οικονομία χαμηλής κατανάλωσης άνθρακα και υψηλή ενεργειακής απόδοσης. Μετά υπήρχε άλλο ένα ερώτημα της κυρίας Μπερμέχο. για το TTIP. Και μετά ρωτήσατε κατά πόσον εμείς ως ε, Σλοβακία είμαστε υπέρ του ο κόσμος, οι πολίτες να αποφασίζουν για, το, για τις ενεργικές υποδομές και το ενεργειακό μείγμα. Είναι σημαντικό θέμα το TTIP και δεν πρέπει το αποτέλεσμα να οδηγήσει σε αποδυνάμωση των ευρωπαϊκών κανόνων, ούτε της υπονόμευσης, να οδηγήσει σε υπονόμευση τη ανταγωνιστικότητας τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά να αξιοποιήσουμε όλε μα τι δυνατότητε. έχοντα κατά νου βεβαίω και του ε, περιορισμού αλλά και τι δυνατότητε που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πρέπει να κινηθούμε βιαστικά κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων σε αυτές τις συμφωνίες. Και νομίζω ότι η ομάδα διαπραγμάτευσης έχει πολλούς τομείς να καλύψει. Πολλά μένουν ακόμα να γίνουν λοιπόν μέχρι την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων. Και για το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, Δηλαδή θα πρέπει οι πολίτες να αποφασίζουν για τις προτεραιότητες τους στον τομέα της ενέργειας. Θεωρώ ότι είναι καλό οι πολίτες ε, να έχουν την δυνατότητα να λαμβάνουν αποφάσεις, εδώ εμπροκειμένου για το ενεργειακό μείγμα, γιατί κάθε χώρα έχει μια ιδιάζουσα κατάσταση με ιδιαίτερες ε, περιστάσεις και συνθήκες. Κάποιες χώρες, ας πούμε, είναι ευνοημένες σε ό,τι αφορά την ηλιακή και ολική ενέργεια. Σε άλλες χώρες ε, υπάρχουν καλύτερες συνθήκες ε, για, την, ε, για να βασίσουν τον ενεργειακό τους μείγμα στην πυρηνική ενέργεια. Αυτή τη στιγμή λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε χώρα παίρνει τις αποφάσεις της ως προς το ενεργειακό της μείγμα. για το καθεστώς ε, οικονομίας αγοράς ε, για την Κίνα. Αναφερθήκατε στο εργατικό δυναμικό στο ερώτημά σας, ήταν πιο συγκεκριμένοι. Όμως, για την χορήγηση αυτού του καθεστώτος στην Κίνα, να σας πω ότι εμείς θα υποστηρίξουμε οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί από κοινού και θα διασφαλίσουμε ότι δεν θα ε, τεθεί ένα αμφιβόλο ούτε θα διακινδυνεύσουμε την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ε, αγοράς. Και το τελευταίο ερώτημα ήταν του κ. Ταμπουράνο. Νομίζω ότι τα κάλυψα όλα όσα είχε θίξει, απαντώντας στους συναδέλφους του. Αν ξέχασα κάτι, ζητώ συγγνώμη και ελπίζω κατά τη διάρκεια των επόμενων ε, μηνών της Σλοβακικής Προεδρίας να έχουμε πολλές ε, ευκαιρίες να εξετάσουμε αυτά τα θέματα, αλλά και διμερώς βεβαίως. Ελπίζω να έχω αρκετό χρόνο να τα συζητήσουμε όλα αυτά, είτε ατύπως, είτε και όχι. Έχουμε και ένα δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Είμαι λοιπόν στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας κύριε Υπουργέ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Ρούμπικ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ, για όλα όσα είπατε. Για μας είναι πάντοτε μεγάλη χαρά να υποδεχόμαστε μια νέα Προεδρία με νέες φιλοδεξίες. Για μας είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε για την διάσκεψη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που σκοπεύετε να διοργανώσετε στην Πρατισλάβα. Θα θέλαμε εμείς να μάθουμε αν σε αυτή τη διάσκεψη θα συζητηθεί και το θέμα της χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων γιατί είναι πολύ, θέμα, ε, πολύ σημαντικό θέμα αυτό στο επόμενο, στην επόμενη ε, περίοδο του προϋπολογισμού. Ε, υπάρχει ο ορίζοντας 2020, ε, υπάρχει το Εράσμους για επιχειρηματίες και υπάρχει και το πρόγραμμα Upscale που έχει ιδιαίτερη σημασία για μας και έχουμε και το Female Business Initial Act όπου προσπαθούμε να προωθήσουμε τη γενική επιχειρηματικότητα. Πιστεύετε ότι αυτά που ανέφερα θα μπορούσαν να είναι θέματα στα οποία θα μπορούσαμε να εμβαθύνουμε ενδεχομένω στο πλαίσιο αυτής της διάσκεψης και η Σλοβακία μήπως θα μπορούσε να θέσει σε προτεραιότητα τα προγράμματα αυτά προκειμένου η υλοποίησή τους να στεφθεί με επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ λέει ο Πρόεδρος, ευχαριστώ για αυτό το ερώτημα. Υπάρχει κάποιος άλλος που θα ήθελε να πάρει το λόγο. Αν μου επιτρέπετε θα ήθελα να προσθέσω και εγώ και να θέσω και εγώ κάποια ερωτήματα. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας κύριε Υπουργέ στο σύστημα εμπορίας εκπομπών. Είναι, είναι βεβαίως ένα θέμα για το οποίο στο Κοινοβούλιο είναι αρμόδια επί της ουσίας η Επιτροπή Περιβάλλοντος. Παρ' όλα αυτά όμως νιώθουμε και εμείς ότι έχουμε μια ανάγκη, ε, ευθύνη ε, απέναντι στις ευρωπαϊκές ε, βιομηχανίες και τις ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό για εμάς το πώς θα μπορέσουμε να ε, αποφύγουμε την διαρροή άνθρακα και τη διαρροή θέσεων εργασίας. Η όλη η συζήτηση λοιπόν που θα γίνει γύρω από αυτό το θέμα θα αποτελέσει προτεραιότητα της, Σλοβακία, της Σλοβακικής Προεδρίας. Ποια είναι λοιπόν η δική σας προσέγγιση από άποψης πολιτικής ενέργειας. Πώς σκοπεύετε εσείς να εμποδίσετε την απώλεια ανταγωνιστικότητας ε, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δεύτερον, για το ζήτημα του, της πράξης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πολύ σημαντικό να μας πείτε ποιες πράξεις θέλετε να, να ε, υλοποιήσετε στην πραγματική οικονομία. Εδώ δεν μιλάμε για μακροοικονομικά στοιχεία, αλλά για τις ε, ευρωπαϊκές βιομηχανίες και τις ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και τρίτο θέμα. Όπως είπε ο ε, συνάδελφος από την ομάδα Γκουε, ενεργειακά ζητήματα και TTIP και σχετικές διαπραγματεύσεις. Γνωρίζουμε ότι οι ενεργειακές τιμές, ιδίως οι τιμές του φυσικού αερίου, στις ε, Ηνωμένε Πολιτείες είναι πολύ χαμηλότερες από ό,τι είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήταν πολύ σημαντικό λοιπόν προτού ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για το TTIP να ανοίξουν τα αμερικανικά σύνορα για τις εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου είναι ένα από τα θέματα που συζητώνται μεταξύ ΙΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποια είναι λοιπόν η στάση της Σλοβακικής Προεδρίας όσον αφορά αυτό το άνοιγμα των ε, εξαγωγών πριν από την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων. Γιατί αν ανοίξουμε τα σύνορα στη βάση του TTIP μεταξύ ΙΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά πάσα πιθανότητα εμείς θα είμαστε χαμένοι όταν υπάρχουν τόσο σημαντικές ε, διαφορές στις ενεργειακές τιμές, ιδίως για τον κλάδο των λοιπασμάτων. Θα ήταν μια καταστροφή λοιπόν. Αυτά είναι τα θέματα που θα ήθελα να θέσω εγώ προς εσάς κύριε Υπουργέ και επειδή δεν βλέπω να υπάρχει κάποιος άλλος που θα ήθελε το λόγο, ε, σας δίνω λοιπόν εσάς το λόγο για να μας απαντήσετε σε αυτές τις τελευταίες παρατηρήσεις που ακούστηκαν. Ε, σας ευχαριστώ πολύ για τις επιπλέον ερωτήσεις που μου υποβάλλατε. Ο κύριος ε, Ρούπικ ε, αναφέρθηκε στο συνέδριο της ε, Μπρατισλάβα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της Σλοβακικής Προεδρίας. Πρέπει να σας πω ότι βεβαίως σας σας ε, προσκαλώ 23 με 25 Νοεμβρίου σε αυτήν την ε, διάσκεψη στόχος της οποίας θα είναι η έγκριση της ε, έκθεσης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για το 2016, ενώ ταυτόχρονα θα ασχοληθούμε με τα γενικότερα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω ε, των εκθέσεων των εισηγητών ενώ θα δώσουμε και ε, τις πιο επικαιροποιημένες πληροφορίες ε, για τον τομέα και βεβαίως θα προετοιμάσει και το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της 28 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες. Η χρηματοδότηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι βεβαίως ένα σημαντικό ζήτημα. Ε, μπορεί να παράσχει ε, χρηματοδότηση μέχρι το 2020 η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω πούμε, του ορίζοντα 2020 ε, που θα μπορούσε να είναι μια πιθανή πηγή επίσης μέσω του προγράμματος COSME. έχουμε την, τον αρμόδιο επιτρόπο που ασχολείται με το θέμα αυτό, όπως επίσης και με την ε, την ε, Κεφαλαϊκή Ένωση και τις ε, κεφαλαιαγορές και τις διαστηνοριακές ε, σχέσεις. Αυτό που μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι θα συνεχίσει η Προεδρία, η Σλοβακική Προεδρία της διαπραγματεύσεις θα ολοκληρώσει το διάλογο όσον αφορά τις συμπράξεις ιδιωτικού δημοσίου καθώς επίσης ε, και όσον αφορά τον ε, ε, κανονισμό για την απλουστευμένη πρόσβαση στις κεφαλαγορές καθώς επίσης και τον κανονισμό Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα απασχολήσει και την άτυπη διάσκεψη της ομάδας Συμμετοπιστωτικών θεμάτων ε, στην Μπρατισλάβα και ε, όλα αυτά λοιπόν θα έχουν σαν στόχο κεντρικό την βελτίωση της κατάστασης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, ο, ο κύριος Πρόεδρος Μπούζεκ υπέβαλε αρκετά ερωτήματα και θα προσπαθήσω να τα απαντήσω όσον αφορά το πρόγραμμα εμπορίας εκπομπών. Οι συνάδελφοι που ασχολούνται με την κλιματική αλλαγή Ε, προτίθενται να δημιουργήσουν τις κατάλληλες ε, συνθήκες έτσι ώστε να προχωρήσουμε ε, προς μια οικονομία πιο αποτελεσματική και που θα χρησιμοποιεί λιγότερο άνθρακα. Ξέρουμε ποιο είναι το πρόγραμμα όσον αφορά την μείωση των εκπομπών μέχρι το 2030. Το προσυπογράφει η Σλοβακική Προεδρία και οπωσδήποτε ε, δεν προτίθεται να αλλάξει ποσοστό στις εθνικές κτλ. Ε, να σας πω πάντως ότι ε, η Σλοβακική Προεδρία διαπραγματεύεται και επιπλέον προτάσεις οι οποίες δεν έχουν αναφερθεί μέχρι τώρα όσον αφορά τις εκπομπές και όσον αφορά την κλιματική αλλαγή. κυρίως ε, δε όσον αφορά τα, το φαινόμενο του θερμοκηπίου και τα αέρια θερμοκηπίου. Όσον αφορά τώρα τη διασφάλιση ίσων ε, ε, ίσων ευκαιριών για την ε, ευρωπαϊκή βιομηχανία και αυτό βεβαίως μας απασχολεί όπως και η σωστή κατανομή των πόρεων, των πόρων κυρίως όσον αφορά τον, την ηλεκτρική ενέργεια και μέχρι το 2030 ευελπιστούμε ε, ότι θα έχει επιτευχθεί αυτή η, αυτό το ε, κοινό ε, επίπεδο και το level playing field όπως το ονομάζουμε στην Ευρώπη. Όσον αφορά τώρα το θέμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις Small Business Act. η δυνατότητα αναθεώρησης ε, του πλαισίου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, και το θέμα το, της δημόσιας διαβούλευσης συζητήθηκε στο Συμβούλιο τον μήνα Δεκέμβριο, καθώς επίσης και του 14 και το Μάιο του 2015. Και αναγγέλθηκε ότι δεν θα υπάρξει αναθεώρηση του εν λόγω πλαισίου και επομένως η Κομισιόν θα συνεχίσει με το ίδιο πλαίσιο του 2011. Εμείς ε, συμφωνούμε απολύτως ως Προεδρία με τις ε, πέντε προτεραιότητες οι οποίες έχουν προκύψει από τις ε, αρχικές διαβουλεύσεις ε, που κύριο γνώμονα έχουν την καλύτερη πρόσβαση ε, των επιχειρήσεων στους, στην χρηματοδότηση καθώς επίσης και στις δυνατότητες κατάρτισης. Ε, εμείς θέλουμε οι προτεραιότητες ε, να μην είναι μόνο λόγια, αλλά να υλοποιηθούν στην πράξη, γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα καλό και αποτελεσματικό πλαίσιο, στο οποίο θα μπορούν να λειτουργούν αποτελεσματικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τέλος, όσον αφορά το άνοιγμα των συνόρων, πριν την ολοκλήρωση της συμφωνίας TTIP, κυρίως όσον αφορά τις εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου. Υπάρχουν βεβαίως πολλά μέτρα τα οποία λαμβάνονται στον τομέα της ενέργειας έτσι ώστε να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει επιτυχώς οποιαδήποτε διακοπή παροχής ε, και ε, ε, εφοδιασμού. Ε, το, η ασφάλεια εφοδιασμού ε, ενέργειας είναι για την Ευρωπαϊκή Ένωση κάτι πάρα πολύ ε, σημαντικό. Και μάλιστα αυτό το έχει, το έχει αναφέρει και ο αρμόδιος ε, επίτροπος. με ρωτήσατε τώρα εάν μπορούμε να συμφωνήσουμε να ανοίξει η αγορά πριν ακόμα και την ολοκλήρωση της ε, TTIP. Σας απαντώ λοιπόν ότι αυτή είναι μια περίπλοκη ερώτηση. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ μονάχα στο υγροποιημένο φυσικό αέριο. γιατί το θέμα του TTIP και των ε, συνθήκων που με την συμφωνία TTIP ε, ε, σχετίζονται είναι ε, ε, ιδιαίτερος περίπλοκο. Απ' την άλλη πλευρά θα πρέπει να μετρήσουμε και τα υπέρ και τα κατά, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα. Ε, και μην λησμονείτε ότι μπορεί, δεν είμαστε μόνο εμείς που μπορεί να έχουμε προβλήματα με την Αμερικανική πλευρά, αλλά και η Αμερικανική πλευρά με μας. Είναι γεγονός ότι η TTIP θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ως ένα ενιαίο πακέτο. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ για την επίσκεψή σας στο ε, ε, Κοινοβούλιο, λέει ο Πρόεδρος Μπούζεκ. θα έχετε ένα εξάμεινο στη διάρκεια του οποίου θα μπορέσετε να επηρεάσετε τα πράγματα και τις συζητήσεις έτσι ώστε να μπορέσετε να προωθήσετε κάποια πράγματα μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους. Σίγουρα η δουλειά σας θα είναι έντονη και ελπίζω και σας εύχομαι να είναι και παραγωγική ε, και ε, περιμένουμε, σας περιμένουμε ε, ξανά. Ναι, ναι, και εγώ βεβαίως ε, ε, προσβλέπω στη συνεργασία με το Κοινοβούλιο, μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για οποιασδήποτε ιδέες προκύψουν από την πλευρά σας, από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ωραία, συνάδελφοι. Ας προχωρήσουμε τώρα στο σημείο 4 της μέσας διάταξης Το λόγο έχει ο κύριος ε, Ρόμαν ε, Βρέτσελη, Υπουργός ε, Μεταφορών, Κατασκευών και Περιφερειακής Ανάπτυξης. μεταφορών δημοσίων έργων λοιπόν ε, και περιφερειακή ανάπτυξη. Ιδίω ό,τι αφορά τα δημόσια έργα ε, θα ήταν ε, με μεγάλο ενδιαφέρον θα σας παρακολουθήσουμε γιατί αυτό συνδέεται ενδεχομένω και με τις τηλεπικοινωνίες. Ξέρουμε ότι ασχολείστε και με το ζητήμα των τηλεπικοινωνιών που είναι πολύ σημαντικό για μας. Παρακαλώ. Καλώς ήρθατε στο Κοινοβούλιο δημόσια έργα, αυτά αφορούν και με την ε, ψήξη και θέρμανση. Και ο συνάδελφός σας προηγουμένως ε, άκουσε πολλά ερωτήματα που άπτονται της ενέργειας, αλλά τώρα θα θέλαμε να επικεντρωθούμε περισσότερο στην πολιτική τηλεπικοινωνιών. Οι φάκελοι τηλεπικοινωνιών ε, με τους οποίους θα καταπιαστεί η ΙΤΡΕ κατά τη διάρκεια της Προεδρίας αφορούν την αναθεώρηση ε, της ε, περιαγωγής χοντρικής, ε, εξαιρετικά σημαντικό θέμα, αναθεώρηση του πακέτου τηλεπικοινωνιών εν γέννη και πρόταση για την ε, χρήση της ζώνης συχνοτήτων 700 MHz. Και να προσθέσω από την αρχή ότι η αναθεώρηση της περιεγωγής χοντρικής φαίνεται ότι είναι εξίσου σημαντικό και επίγον ζήτημα όπως και στην περίπτωση της ε, ασφάλειας εφοδιασμού φυσικού αερίου. Για την Επιτροπή μας λοιπόν και τα δύο ζητήματα είναι κέρια σημασίας και τα εξετάζουμε ως επίγοντα και το τονίζω αυτό. Θα θέλαμε να οριστικοποιηθούν και τα δύο αυτά θέματα κατά τη διάρκεια της Προεδρίας. Και τα δύο. Αυτά τα δύο που προανέφερα. Αν θέλουμε να μην υπάρχουν πλέον τέλη περιαγωγής μέχρι τον επόμενο Ιούνιο. Ωραία, παρακαλώ, έχετε το λόγο, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ. Όλα έχουν ήδη υποθεί βεβαίω από τον συνάδελφο που παρουσίασε τους ε, στόχους και τις προτεραιότητες μας. Παρ' όλα αυτά, να χαιρετήσω επισήμω και εσά, κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίε και κύριοι. Είναι μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι εδώ σήμερα και να σα παρουσιάσω τι ε, προτεραιότητε τη Λογική Προεδρία ε, στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αλλά και για το πρόγραμμα Γαλιλαίου. Όπως φαντάζεστε, η 1η Ιουλίου ήταν ε, μία πρωτοφανής ημέρα για μας. Τώρα ξεκινάνε ε, οι εργασίες μας. Για πρώτη φορά έχουμε αναλάβει την εκπαιδευτική προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα σε δύσκολες ε, συνθήκες δεδομένων των πρόσφατων εξελίξεων. Παρ' όλα αυτά, είμαστε πανέτοιμοι να συνεχίσουμε τις ε, προσπάθειες και να τέθουμε επικεφαλή των συζητήσεων κατά τη διάρκεια του επόμενου εξαμήνου. Σε στενή βεβαίω συνεργασία με τους συναδέλφους ε, του Τρίτου Προεδριών, σε αγαστή συνεργασία και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ενίσχυση της ε, ενιαίας ψηφιακής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά θα ήθελα να πείτε και εσείς ποιες είναι οι δικές σας ε, προτεραιότητες, ποια είναι τα κύρια για σας ζητήματα και πώς μπορούμε να βρούμε ε, τρόπους βελτίωσης ε, του έργου μας στο Συμβούλιο αλλά και ενίσχυσης της αμοιβαίας αυτής της συνεργασίας οι επικοινωνικές σχέσεις μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων που είναι και συνομοθέτε από κοινού και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι απαραίτητη προπόθεση αν θέλουμε να επιτύχουμε αυτά αποτελέσματα και να αποφύγουμε τον κατακαιρματισμό της εσωτερικής αγοράς. Ιδιαιτέρως μετά τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξει ε, βλέπουμε ότι υπάρχει πραγματική πρόκληση ε, για τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει λοιπόν το αποτέλεσμα του Βρετανικού Δημοψηφίσματος ε, να μας οδηγήσει ε, στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε ε, μεγαλύτερες και βαθύτερες συνδέσεις με τους Ευρωπαίους πολίτες, μεγαλύτερη διαφάνεια και ότι θα πρέπει να διαμορφώσουμε τις προϋποθέσεις για τις επιχειρήσεις, τις μικροπιστές επιχειρήσεις και τους πολίτες γενικότερα. Εμείς ε, αυτό θέτουμε ως κύριο γνώμονα για την Προεδρία μας για το επόμενο εξάμεινο προκειμένου να βελτιώσουμε με πολύ απτό τρόπο τις ζωές των Ευρωπαίων πολιτών. Σε στενή συνεργασία με τους συναδέλφους από την Τριάδα των ε, Προεδριών θα εργαστούμε επισταμένως για την υλοποίηση της, ε, της στρατηγικής για την ενιαία ψηφιακή αγορά που υιοθετήθηκε πέρσι τέτοια εποχή είναι μια καλή ευκαιρία να αξιολογήσουμε και να κάνουμε έναν απολογισμό τη σημερινή κατάσταση ω προ τη στρατηγική αυτή και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Εξετάζουμε λοιπόν ε, την ε, ενιαία ψηφιακή αγορά ω μια μοναδική ευκαιρία και για την οικονομία αλλά και για ένα θετικό θεματολόγιο που εξυπηρετεί του στόχου του κοινού μα ευρωπαϊκού εγχειρήματο. Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και τη τεχνολογία πληροφοριών, η Σλοβακική Δημοκρατία χαιρετίζει την υιοθέτηση υπό Ολλανδική Προεδρία τη Γενική Προσέγγιση για την πρόταση εναρμόνιση τη ζώνη συχνοτήτων 700 MHz. Αυτό το επίτευγμα επιτρέπει στη Σλοβική κυβέρνηση, στην Προεδρία, να ξεκινήσει διαπραγματεύσει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτός ο φάκελος. Η νομοθεσία αυτή είναι απαραίτητη όχι μόνο για να διαμορφώσει το έδαφος για την ανάπτυξη των υπηρεσιών 5, 5G, αλλά και για να διατηρήσουμε το χαμηλότερο μέρος ε, του εύρου συχνοτήτων UHF ε, για την επίγεια παροχή ε, υπηρεσιών εκπομπών με την δωρεάν τηλεόραση, για την χρήση του ασύρματου ε, ακουστικού προγράμματος και ούτω καθεξής. Αναγνωρίζουμε ότι είναι σημαντική προθεσμία του 2020, αλλά θα πρέπει να έχουμε και ένα περιθώριο ευελιξίας, καθώς η τροποποίηση ε, της εκπομπής τηλεοπτικών δικτύων μπορεί να είναι κάτι δαπανηρό, αλλά και χρονοβόρο. Από ό,τι βλέπω, δεν ε, υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου για αυτό το θέμα. Γι' αυτό προσβλέπω σε αγαστή συνεργασία και σε επίτευξη συμφωνία για αυτό το φάκελο. Η Σλοβακική κυβέρνηση θα ε, καταβάλει κάθε προσπάθεια για την ε, διασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατή προόδου διαπραγματεύσει για την αναθεώρηση της περιαγωγή χονδρικής, το οποίο αποτελεί απαραίτητη προπόθεση για την κατάργηση των τελών περιαγωγή από τον Ιούνιο του 2017 και μετά. Η επιτυχής ε, ολοκλήρωση αυτών των διαπραγματεύσεων θα αποτελέσει ε, μεγάλη νίκη και επίτευγμα για τους καταναλωτές, αλλά και μεγάλο βήμα προς ε, την ενιαία ψηφιακή αγορά στην Ευρώπη. Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ως συνομοθέτες πρέπει να επιτύχουν συμφωνία μέχρι το Φεβρουάριο του 2017, προκειμένου να υλοποιηθεί αυτός ο στόχος. Γι' αυτό το λόγο βασιζόμαστε στη δική σας ε, προθυμία και την ετοιμότητά σας να ξεκινήσουν πραγματεύσει το συντομότερο δυνατό. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εξεύρουμε έναν επικοδομητικό συμβιβασμό στα ζητήματα που εκκρεμούν. Μια άλλη σημαντική νομική πράξη που είναι ε, ουσιαστική σημασία για τη δημιουργία της ψηφιακή ενιαίας αγορά είναι η αναθεώρηση του ρυθμιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, τα δίκτυα και τις σχετικές υπηρεσίε που θα παρουσιαστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά το καλοκαίρι. Ο εξυγχρονισμό του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις τηλεπικοινωνίες είναι αναπόφευκτος λόγω της αύξησης της ζήτησης ε, για υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων, την, ε, το χάσμα μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών όσον αφορά τα ψηφιακά ζητήματα που εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά και τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, τους νέους φορείς, τους νέους παίκτες στην ε, αγορά των online υπηρεσιών. Η Σλοβακική Προεδρία θα ε, ηγηθεί μιας πολιτικής συζήτησης που θα γίνει ε, ε, επί των στοιχείων της αναθεώρησης κατά την διάρκεια του Συμβουλίου για τις Τελεπικοινωνίες που θα γίνει στις 2 Δεκεμβρίου φέτος και θα προετοιμάσει το έδαφος για τα θέματα αυτά για την Μαλτεζική Προεδρία. Τέλος, να αναφερθώ και στο ζήτημα του GNSS, του Παγκόσμιου Δορυφορικού Συστήματος Πλοήγησης και πιο συγκεκριμένα του, για το Γαλιλαίο. Το 16 αποτελεί σημαντικότατο ορόσημο στην ανάπτυξη του προγράμματος Γαλιλαίου. Αυτόν τον χρόνο, φέτος δηλαδή, θα δούμε να ξεκινούν οι πρώτες αρχικές υπηρεσίες που παρέχουν τα σήματα Γαλιλαίου. Και ως ε, χώρα που κατέχει τη θέση της Προεδρίας, εμείς θέλουμε να ενστερνιστούμε την στρατηγική που έχει χαραχτεί στον τομέα αυτό, τον, ε, τον, τη στρατηγική για, την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το διάστημα. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρξουν νέες επενδύσεις στον τομέα των εφαρμογών, κάτι που θα επιφέρει κοινωνικά και οικονομικά ωφέλη. Θα θέλαμε επίσης για άλλη μία φορά να επιβεβαιώσουμε από την δική μας πλευρά την ετοιμότητά μας να συνεχίσουμε τις κοινέ ευρωπαϊκές προσπάθειες προκειμένου το Γαλιλαίο να καταστεί λειτουργικό, πλήρως λειτουργικό έως το 2020. Αγαπητά μέλη, αυτές είναι οι προτεραιότητες μας στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και της ε, παγκόσμιας δορυφορικής πλοήγησης. Βασίζομαι στη δική σας υποστήριξη και πιστεύω ότι θα επιτύχουμε πολύ θετικά αποτελέσματα με όφελος για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Ανυπομονώ λοιπόν να συνεργαστούμε και είμαι στη διάθεσή σας για οποιασδήποτε ερωτήσεις έχετε. Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους των πολιτικών ομάδων, λέει ο Πρόεδρος, πρώτα απ' όλα η κυρία Δελκαστήριο Βέρ, που είναι η συγγήτριά μας για τη δέσμη ε, για τις τηλεπικοινωνίες, εκ μέρους του ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ε, καλωσορίζω κύριε Υπουργέ και εγώ από την πλευρά μας στον τομέα της ψηφιακής ε, μεταμόρφωσης πραγματικά αντιμετωπίζουμε μια πραγματική επανάσταση και αποτελεί το θέμα αυτό ε, σημαντικό θέμα για την ευρωπαϊκή οικονομία. Αν δεν ψηφιοποιηθούμε, η ευρωπαϊκή οικονομία δεν θα έχει τους επαρκείς και απαραίτητους ε, πόρους προκειμένου να ηγηθεί των παγκόσμιων αγορών. Άρα αυτό το θέμα πραγματικά άπτεται της ανάπτυξης του, της, ε, του ψηφιακού τομέα της οικονομίας μας. Αναφερθήκατε στις τέσσερις διαστάσεις αυτής της πολιτικής ε, που έχετε σκοπό να υλοποιήσετε ε, με αφορμή την ανάληψη των καθηκόντων σας. Θα ήθελα ωστόσο να επικεντρωθώ σε μία από τις διαστάσεις που από άποψη χρόνου είναι η πιο επίγουσα, που είναι η αναθεώρηση της αγοράς ε, χονδρικής. Έχουμε δεσμευτεί τα τρία θεσμικά όργανα να τηρήσουμε μια συγκεκριμένη προθεσμία. Και θα ήταν καταστροφή για τους Ευρωπαίους πολίτες, αν δεν τα καταφέρουμε να την τηρήσουμε, που είναι το τέλος των χρεώσεων περιαγωγής από τα μέσα Ιουνίου του 2017. Και από αυτή την άποψη πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό πώς εσείς θα μπορούσατε να επιταχύνετε την όλη διαδικασία προκειμένου να επιτύχουμε τον συγκεκριμένο στόχο και να καταλήξει το Συμβούλιο σε ε, οριστική θέση προκειμένου να ξεκινήσουν και οι διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο. Δεύτερο θέμα. Θα ήθελα να αναφερθώ στο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις τηλεπικοινωνίες και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Αυτό αυτή τη στιγμή δεν, δεν συζητείται ακόμα, γιατί η πρόταση της Κομισιόν δεν έχει κατατεθεί ακόμα. Θα γίνει βέβαια το Σεπτέμβριο, αλλά ε, Ούτε εμεί ω κοινοβούλιο δεν θα είμαστε έτοιμοι μέχρι το τέλος του χρόνου. Αλλά πρόκειται για ένα θέμα το οποίο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό όχι μόνο από το τι θα κάνει η Προεδρία, μπορεί να χρειαστεί και άλλη μία Προεδρία ή και άλλη μία, αλλά εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από το τι έχει ήδη γίνει από τις δύο προηγούμενες Προεδρίες. Γιατί έχετε, κατά τη γνώμη μου, το Συμβούλιο θα πρέπει αμέσως μετά την υποβολή της πρότασης από την Κομισιόν, ε, το Συμβούλιο λοιπόν θα πρέπει αμέσως να ξεκινήσει τις εσωτερικές του συζητήσεις, γιατί αν δεν το κάνει θα είναι αδύνατον να ολοκληρωθούν αυτές οι συζητήσεις εντός δύο ετών. Μπορεί να χρειαστούν πολύ περισσότερα χρόνια. Θα ήθελα λοιπόν να σας ασκήσω μια κάποια πίεση και βεβαίω είμαι σίγουρη ότι έχετε την πολιτική βούληση. Αλλά θα ήθελα και εγώ άλλη μια φορά να σας το πω. Μόλις η Κομισιόν δημοσιεύσει την πρότασή τη για την αναθεώρηση του ρυθμιστικού πλαισίου για τις τηλεπικοινωνίες και τις ηλεκτρονικέ επικοινωνίες είναι πάρα πολύ σημαντικό εσείς από τη θέση τη Προεδρία να ξεκινήσετε συζητήσει στο Συμβούλιο γιατί αν δεν το κάνετε δεν θα καταλήξουμε ενδεχομένως ούτε καν ε, μέχρι το τέλος της κοινοβουλευτικής αυτής θητείας. Και αυτό θα είναι καταστροφή. Η Ευρώπη χρειάζεται τις κατάλληλες απαντήσεις τον κατάλληλο χρόνο στα σημαντικά ερωτήματα. Και αυτό το ζήτημα που σχετίζεται με το, ρυθμιστικό, με το ρυθμιστικό πλαίσιο είναι ένα από αυτά τα πολύ ουσιώδη ζητήματα. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Τώρα θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον κύριο Τονασόφσκι εκ μέρου του ECR. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω τσεχικά. Χαίρομαι πολύ που ήρθατε τόσο γρήγορα στην δική μας επιτροπή και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για όλα όσα είπατε σχετικά με τις τηλεπικοινωνίες και τα συστήματα δορυφορικής πλοήγησης. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα θέματα ε, και θα μας απασχολήσουν το επόμενο εξάμεινο σοβαρά. Όσον αφορά τον Γαλιλαίο, έχω ένα ερώτημα να σας θέσω. Αναγνωρίζω ότι τονίσατε τη σημασία του συστήματος Γαλιλαίου και GNSS. Μήπως θα μπορούσατε στη διάρκεια της Προεδρίας σας να επιταχύνετε τις δραστηριότητες σας στον τομέα του GNSS, όπως για παράδειγμα και στο θέμα των ε, διοδίων, όπου η Σλοβακία είναι μια χώρα εξαιρετικά προηγμένη για το πώς θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν δηλαδή αυτά τα συστήματα ή και στο θέμα της παραγωγής των chipset στο Γαλιλαίο. Πρόκειται για ένα πανευρωπαϊκό πρόγραμμα και χρειάζεται να είναι διαθέσιμες σε όλους τους πολίτες και σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς όλες οι πληροφορίες. Χαίρομαι επίσης και για αυτό που είπατε για την κατάργηση των χρεώσεων περιαγωγής. Το ερώτημά μου είναι, θεωρείτε ότι θα υπάρξει πρόβλημα, προβλέπετε ότι θα υπάρξουν προβλήματα όσον αφορά την τήρηση της προθεσμίας που έχει τεθεί του Ιουνίου του 2017. Γιατί εμείς πρέπει να σας πω ότι ελπίζουμε να τηρηθεί η συγκεκριμένη προθεσμία. Το ερώτημά μου είναι αν εσείς πιστεύετε ότι ενδεχομένως θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα ως προς την τήρηση αυτής της προθεσμίας. Κατά τα άλλα, ε, σας διαβεβαιώ από την πλευρά μου και από την πλευρά της Επιτροπής ότι θα είμαστε στη διάθεσή σας για συνεργασία. Η κυρία ε, Κάλες, Κα, από την Άλντε που είναι η συγγήτρια για την ψηφιακή ενιαία αγορά. Μια πολύ απλή ερώτηση έχω, αλλά και πολύ ανοιχτή ερώτηση για την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας και της ε, ε, βιομηχανίας και της ε, οικονομίας ε, χρειαζόμαστε συνδεσιμότητα. Ε, τι θα κάνει λοιπόν η Σλοβική Προεδρία για την οικοδόμηση δικτύων, θα επενδύσει στα δίκτυα, πώς θα αντιμετωπίσει το θέμα αυτό. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρος. Έχουμε και άλλο ένα αίτημα από την πλευρά του κυρίου Ρούμπικ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. το ζήτημα της ε, περιαγωγής χονδρικής ε, για μας είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα όσον αφορά τη δημιουργία και την ε, θέσπιση της ψηφιακής ενίας αγοράς. Και θεωρούμε ότι όλες οι εταιρείες στην Ευρώπη θα πρέπει με διαφάνεια και να προσέρχονται στον ανταγωνισμό και γι' αυτόν τον λόγο το ουσιώδες ερώτημα που ανακύπτει είναι το εξή. Η πρόταση της Κομισιόν είναι ολοκληρωμένη σίγουρα, αλλά μήπως θα, συμφωνήσατε, συμφωνούσατε κι εσείς ότι στο μέλλον θα ήταν καλό να υπάρξει ένα χρηματιστήριο τεραμπάιτ και γιγκαμπάιτ πανευρωπαϊκού χαρακτήρα, προκειμένου να δημιουργηθεί μια πραγματική ενιαία ψηφιακή αγορά. Δεύτερον, εναρμόνιση των συχνοτήτων που είναι απολύτως απαραίτητη για την ανάπτυξη των υπηρεσιών πέμπτης γενιάς. Πιστεύετε ότι υφίσταται ήδη το, ε, υπάρχ, υφίσταται ήδη το αναγκαίο πλαίσιο για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ε, από την δημοπρασία που έχει ε, διοργανωθεί, έχει προγραμματιστεί, θα, έχ, θα διατεθούν τα αναγκαία κεφάλαια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προκειμένου να εξασφαλιστεί ε, η παροχή αυτών των ε, υπηρεσιών 5G. Εμείς σε σχέση με την Ιαπωνία και την Νότιο Κορέα ε, βρισκόμαστε ήδη δύο χρόνια πίσω γιατί οι χώρες αυτές έχουν θέσει ως στόχο να αναπτύξουν το σύστημά τους το 2018 ενώ εμείς το 2020 και επίσης θα θέλω να μου πείτε για το ζήτημα των ε, οπτικών ινών. Ευχαριστώ πολύ λέει, κυρία Κούνε. Είστε και υπεύθυνο για τι μεταφορές και αύριο θα, έρθει, θα ε, εμφανιστείτε ενώπιον της Επιτροπής ε, Μεταφορών. Ξέρετε ποιο, πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν οι μεταφορές ε, και για την Οικονομική αλλά και την ελληνική Ένωσή μα. Και γνωρίζουμε ότι και η Κομισιόν θα, επόμενε εβδομάδε εβδομάδες θα προχωρήσει σε δημοσίευση ανακοίνωση όσον αφορά την, την μείωση του άνθρακα όσον αφορά τι ευρωπαϊκέ μεταφορέ. Έχετε κάτι πιο συγκεκριμένο να μας πείτε γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω κι εγώ από τη δικιά μου πλευρά δύο ερωτήματα στα ε, σχόλια τα οποία ακούστηκαν μέχρι τώρα. Σας ρωτώ, ως Σλοβική Προεδρία είστε έτοιμος να προχωρήσετε το θέμα του ευρωπαϊκού φάσματος πέρα εκτός από τα 700 MHz γιατί το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι απολύτως προφανές ότι τα κράτη-μέλη δεν είναι φύλλα προσκύμενα σε δημιουργία αυτού του φάσματος σε γενικές γραμμές. Δεύτερον, την άποψή σας θα ήθελα όσον αφορά τη δημιουργία βιομηχανικών πλατφορμών δηλαδή τη δυνατότητα ε, να χρησιμοποιηθεί η βιομηχανία ε, για τη δημιουργία ε, πλατφορμών For German industry, ε, γιατί καταλαβαίνετε ότι ε, λαμβάνοντας υπόψη και τις σχέσεις μας με τις ΗΠΑ θα πρέπει να δημιουργηθούν ε, τάχιστα τέτοιου είδους ε, πλατφόρμες. Είχαμε μάλιστα και μία σχετική ακρόαση στην Επιτροπή μας ε, για αυτές τις .zero platforms και την ευρωπαϊκή τους διάσταση. Εσείς πώς βλέπετε τα θέματα αυτά το θέμα του φάσματος δηλαδή, του γενικού φάσματος και της ε, δημιουργίας των βιομηχανικών πλατφορμών κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας. Πώς θα τα αντιμετωπίσετε τα θέματα αυτά. Στρέφομαι τώρα και προς τους συναδέλφους. Θέλει κάποιος να πάρει το λόγο, θέλει να υποβάλει κάποιο ερώτημα, όχι. Αυτές είναι οι ερωτήσεις μας λοιπόν κύριε Υπουργέ, παρακαλώ έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω λοιπόν να απαντήσω. Πρώτα μια ερώτηση τη κυρία Τελκαστήγιο σχετικά για την περιαγωγή. Ε, κοιτάξτε, το μεγαλύτερο ζήτημα εδώ είναι η ταχύτητα. Νομίζω ότι τώρα έχουμε τη μοναδική ευκαιρία στη διάρκεια της Προεδρίας μας ε, να κλείσουμε το θέμα αυτό, να γίνει η συμφωνία. Δεν είναι βεβαίως ε, εύκολο θέμα, αλλά και δεν είναι εύκολο να βρούμε έτσι, τους κοινούς παρανομαστές με όλες τις ε, χώρες όσον αφορά μια κοινή αντίληψη δηλαδή για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα των επιπλέον χρεώσεων στο θέμα αυτό τις ε, περιαγωγές. Ε, περιαγωγές. Επομένως, συζητήσεις ε, θα γίνουν έτσι ώστε να βρεθεί ένα, μια λύση η οποία θα είναι δίκαιη για όλους τους εμπλεκόμενους. Ρυθμιστικό πλαίσιο. το Συμβούλιο είναι γεγονός ότι ε, προσπαθεί να ε, δημιουργήσει τις ε, κατάλληλες προϋποθέσεις και συνθήκες για αυτές τις υπηρεσίες και βεβαίως επικεντρωνόμενο κυρίως στις ανάγκες συνδεσιμότητας. Αυτή είναι η απάντηση, αλλά πώς να σας το πω, θα πρέπει να το ξαναδούμε το θέμα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο, γιατί στενά είναι συνδεδεμένο το ζήτημα αυτό με την εναρμόνιση των ε, συχνοτήτων και με την ενιαία ψηφιακή αγορά και αν θέλουμε πραγματικά να είμαστε σύμφωνοι με την εποχή μας θα πρέπει να τα συζητήσουμε και να τα προχωρήσουμε τα θέματα αυτά. Μια ερώτηση του κ. Τοσινόφσκι. What Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα με την περιαγωγή. Είναι σημαντικό μας μας, σας το είπα και προηγουμένως, προσπαθούμε να βρούμε την καλύτερη δυνατή ισορροπία όσον αφορά το θέμα αυτό. Γιατί από τη μία πλευρά θέλουμε ε, να έχουν την δυνατότητα να είναι αρκετά χαμηλά δηλαδή τα τέλη έτσι ώστε ε, να μπορούν οι εταιρείε ε, να παρέχουν τις υπηρεσίες που πρέπει και στο εξωτερικό αλλά και από την άλλη πλευρά να είναι αρκετά υψηλά έτσι ώστε να μπορέσουν να παραμείνουν οι παίκτες στην αγορά. Δεν είναι απλά πράγματα αυτά. Ξέρετε Ξέρετε ότι ε, μέχρι τώρα είχαμε το 0,5 MB, τώρα η χρέωση προτείνεται να είναι 0,85. Θα δούμε. Uh, was also from Mr. Επίσης, άλλη ερώτηση του κ. όσον αφορά τον Γαλιλαίο. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι ο Γαλιλαίος είναι ευκαιρία, έτσι τον βλέπω εγώ, μια ευκαιρία και για επενδύσεις, ευκαιρία ανεξάρτηση, ανεξαρτητοποίησης από το GSM. Και οπωσδήποτε εγώ βλέπω το θέμα αυτό ενταγμένο και στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Διαστήματος. Και να σας πω ότι εμείς δουλεύουμε ήδη και σε ένα πρόγραμμα συλλογική που θα μπορούσε να αποτελέσει έτσι οδηγό. Τι άλλο με έχετε ρωτήσει για να δω τα χαρτιά μου. Ναι, για την περιέγωγη τα είπαμε ήδη, να μην τα ξαναλέμε. Okay, Madam there was the uh, investments. Uh, and high network will definitely require uh, ε, τώρα όλα αυτά βεβαίως ε, χρειάζονται ε, πολλές ε, επενδύσεις, αλλά αυτό είναι συνθήκη εκ των όνου κάνευ. Αν θέλουμε να προχωρήσει και η, πέμπτη, η συνδεσιμότητα πέμπτης γενιάς για τη βιομηχανία, για τα διασυνδεμένα αυτοκίνητα, όλα αυτά είναι, περνάνε οπωσδήποτε από την καλύτερη συναισθηματικότητα. Τι να λέμε τώρα, έτσι είναι. Άλλο, ναι, μικρότερη, ή λιγότερη χρήση άνθρακα. Αυτό είναι το αγαπημένο μου θέμα και τι σχετίζεται και με τις μεταφορές και είναι και ε, μία από τις ε, κύριες προτεραιότητες τις οποίες ε, θα έχουμε. Η προσέγγιση μας όσον αφορά το θέμα αυτό είναι πολύ σοβαρή και θεωρούμε ότι αυτό το θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό και με μεγάλη βαρύτητα για το μέλλον γιατί, γιατί το 70% των εκπομπών στις περισσότερες χώρες ε, αντιπροσωπεύεται από, το... από, τις, ε, βιο... από τις μεταφορές και στο θέμα βεβαίως των αεροπορικών μεταφορών η προσέγγιση αυτή ε, της ε, ε, ε του άνθρακα, όπως άλλωστε και στην αυσιπλοεία, είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Και επομένως... Ε, ε, πρέπει κάτι να κάνουμε. Ε, οπωσδήποτε θέλουμε και ε, να δώσουμε κίνητρα στον κόσμο να σταματήσει να παίρνει το αυτοκίνητό του, να χρησιμοποιήσει ας πούμε αυτοκίνητα και συγγνώμη, το ποδήλατό του αντί για το αυτοκίνητό του, να παίρνει το τρένο αντί για το μεμονωμένο αυτοκίνητο. Ε, να αλλάξει δηλαδή τον τρόπο της ε, κινητικότητάς του, ε, να κινητροδοτήσουμε τον κόσμο έτσι ώστε να αλλάξει νοοτροπία. Αυτό βεβαίως προϋποθέτει και αλλαγή συνηθιών οι οποίες προκύπτουν μέσα από διδασκαλία, μέσα από εκπαίδευση, μέσα από προσπάθεια. Ε, γιατί καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι μπορεί να φρημάρει αν έχει χρησιμοποιεί μία BMW με άπειρα άλογα μέσα σε μια πόλη, αλλά ότι αυτό μπορεί να είναι πολύ κακό για το περιβάλλον, άρα πρέπει να αλλάξει ε, η νοοτροπία, πρέπει να αλλάξει η παιδεία να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε τις μεταφορές και τις μετακινήσεις μας. Ευχαριστώ πολύ. Α, έχω και κάτι άλλο, ναι. Ποια άλλη ερώτηση. Yeah, what was what are our plans regarding the debate on online platforms, collaborative economy, we support. Συνεργατική οικονομία, πλατφόρμες. Ε, αυτά είναι πράγματα τώρα που είναι πολύ σημαντικά όσον αφορά την ε, οικονομία μας, την τωρινή. Τα ξέρουμε, πρέπει να προχωρήσουμε, γιατί καταλαβαίνετε ότι πρέπει να υπάρξουν ε, ρήξεις όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο ε, βλέπουμε την οικονομία. Πρέπει να δώσουμε ε, μια νέα ροπή επαναστατική στην οικονομία. Επίσης θα πρέπει να ξαναδούμε τον τρόπο με τον οποίο συλλέγονται και χρησιμοποιούνται τα δεδομένα, θα πρέπει να έχουμε ε, διασφάλιση του περιεχομένου κτλ. Γι' αυτό ε, καλούμε άλλωστε και την ε, Επιτροπή να προχωρήσει το ζήτημα των πλατφορμών, των επιγραμμικών online platforms. What was Είσαστε έτοιμοι, ε, Σλοβακική Προεδρία, να πιέσετε το Συμβούλιο προς, ε, το, προς την πολιτική του ευρωπαϊκού φάσματος και αυτό το ζήτημα των 700 MHz. Αυτό είναι, μας ενδιαφέρει πολύ. Δεν είναι εύκολο να υπάρχει ξεκινή προσέγγιση, αλλά είσαστε έτοιμοι, ναι ή όχι. Ναι, είμαστε έτοιμοι είναι η απάντηση. Και θεωρούμε ότι είναι, όπως είπα και προηγουμένως, προϋπόθεση εκ των όνου κάνευ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, σας ευχαριστούμε για τις απαντήσεις σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την δέσμευση την οποία έχετε αναλάβει. Σας ευχόμαστε τα καλύτερα για τη διάρκεια την εξάμηνη της Προεδρίας σας. Μεθαύριο θα είμαστε στην Πρατισλάβα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας να είμαστε ε, παρόντες στην Σλοβακία στη διάρκεια ε, της ε, Προεδρίας της χώρας αυτής. Θα είμαστε μία πρώτη φορά στην Πρατισλάβα, στη Σλοβακία, εν πάση περιπτώσει τον Ιούλιο, άλλη μία φορά το Σεπτέμβριο και έπεται συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λέει και ο κύριος Μπρεσέλη Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζει ο Πρόεδρος. Προχωράμε στο σημείο 5. Νέα στρατηγική για το υγροποιημένο φυσικό αέριο και την αποθήκευση του αερίου. LNG λοιπόν, στρατηγική για το υγροποιημένο αέριο από της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ε, αυτό είναι μέρος του Winter Package, όπως γνωρίζετε ο συνάδελφος που είναι υπεύθυνο για το θέμα αυτό και είναι εισηγητή είναι ο Ανδρέας Γκιούρκ. Αγαπητέ συνάδελφε, μπορείτε να πάρετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που υπέβαλαν τροπολογίες και συνέβαλαν στην έκθεση. Έλαβα 265 τροπολογίες που εκπροσωπούν ένα ευρύ φάσμα ε, απόψεων. Παρ' όλα αυτά τα καταφέραμε και νομίζω ότι έτσι έχουμε μια πλήρη έκθεση και με τις συμβολή των ε, και μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα πλήρες ε, πλαίσιο. Βασίστηκα σε τρεις ε, αρχές για την εκπόνηση της έκθεσης αυτής. στόχος και στόχευση, ισορροπία και εκπροσώπευση. Ήθελα λοιπόν να επικεντρωθούμε ε, ακριβώ στο ζήτημα το οποίο μα απασχολεί. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Δεν θέλαμε να το παραφορτώσουμε και να βάλουμε οποιοδήποτε θέμα κάποιο θεωρεί ότι έχει την ελάχιστη σύνδεση με αυτό το ζήτημα. Γιατί αυτό θα ε, περιέπλεκε τα πράγματα και θα επαναρχόμασταν ε, στην αφετηρία μα ω προ την Ενεργειακή Ένωση ή θα προσπαθούσαμε από την άλλη να προβλέψουμε οποιαδήποτε οποιοδήποτε υποσενάριο εκ των προτέρων. Θέλουμε λοιπόν να επικεντρωθούμε στη, στα ζητήματα ουσία. Η στρατηγική είναι πιο σημαντική για ορισμένα κρατημέλη. Υπάρχει και γεωγραφική διάσταση δηλαδή. Αυτό είναι αναμφίβολο. Ε, κάποιοι έχουν ε, έξι ε, τέτοιου ε, σταθμού φυσικού αερίου, κάποιοι καθόλου. Κάποιοι μπορούν να καλύψουν κατά 100% τι ανάγκε στο φυσικό αέριο, κάποιοι καθόλου. Ε, και αυτό θα έπρεπε να διαμορφώσει τελικά μία λύση που να ικανοποιεί του πάντε. Θέλαμε λοιπόν να υπάρχει ισορροπία για του επιμέρου ε, στόχου, για την διασφάλιση τη ασφάλεια εφοδιασμού, την προώθηση τη βιωσιμότητα ε, και την προώθηση τη ανταγωνιστικότητα με προσιτέ τιμέ. Και οι τρει αυτοί στόχοι θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται για να έχουμε μια καλή ε, έκθεση. Η τρίτη αρχή που ακολούθησα ήταν να είναι αντιπροσωπευτική η έκθεση για το σύνολο του Κοινοβουλίου ή δυνατόν. Και ρίμνησα τους ώστε όλες οι ε, τροπολογίες όλων των πολιτικών ομάδων να λαμβάνονται υπόψη. Τελικά αξιοποίησα το 1 τρίτο των ε, τροπολογιών στις συμβαστικές τροπολογίες μου και νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτή η έκθεση να έχει όσο το δυνατόν ευρύτερη στήριξη από το Κοινοβούλιο. Κατά τη γνώμη μου, αυτοί οι τρει στόχοι είναι προφανώ ανηλέντετοι. Αυτή η έκθεση μπορεί να τύχει ευρύτερη στήριξη μόνο αν είναι και ισορροπημένη αλλά και στοχευμένη. Επομένω, είναι προ το συμφέρον όλων να δείξουμε ότι υπάρχει ευρεία στήριξη γιατί ε, όταν είμαστε ενωμένοι έχει και η φωνή μα μεγαλύτερη ισχύ. Πρέπει λοιπόν να ε, λύσουμε εσωτερικά τις ε, διαφορές μας ε, και να μιλήσουμε με ενιαία φωνή ή δυνατόν. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι, ιδίως τους σκιώδεις συζητητές και προβλέπω σε συνέχιση των κοινών μας εργασιών. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφε για τα σχολιά σου. Το λόγο έχουν τώρα οι σκιώδεις από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες ο συνάδελφος ε, Γανονάτο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή Ανδρέα Γκιούρκ για τις διαπραγματεύσεις που έκανε με εξαιρετική διάθεση συμφιλίωσης και πνεύμα συνεργασίας έτσι ώστε να βρεθεί ένα καλό κείμενο το οποίο να μπορεί ε, να ε, υποστηριχθεί από την πλειοψηφία. Ε, βλέπω τις τροπολογίες και θεωρώ ότι θα πρέπει να βρεθεί κάποια σύνθεση μεταξύ των διαφόρων τροπολογιών που πολλές είναι ταυτόσιμες. Ε, θεωρώ ότι κυρίως θα πρέπει να ασχοληθούμε με τον μακροπρόθεσμο στόχο της ε, ε, μείωσης της χρήσης του άνθρακα, καθώς επίσης τη μείωση της εξάρτησης από, τις, τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Αυτό είναι μια πρακτική, μια πολιτική η οποία θα πρέπει να συνεχιστεί με τρόπο ώστε να υπάρχει σύγκληση με τους στόχους για το 2050. Επίσης, ε, θεωρούμε ότι θα πρέπει να ε, αναφερθεί η καλή χρήση ε, των υφισταμένων υποδομών. Είναι κοινό τόπος και συμφωνούν όλοι από αυτού ότι υποχρησιμοποιούνται οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις. Ε, επίσης, ε, όσον αφορά τους χερσαίους διαδρόμους ε, βορρά-νότου Ανατολής-Δύσης, θα πρέπει ιδιαίτερως να προσεχθούν οι πιο επικίνδυνες χώρες. Όσον αφορά ε, την χρήση ε, του υγροποιημένου αερίου στις μεταφορές ως εναλλακτικού ε, καυσίμου πιστεύω ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να προτιμηθεί σε σχέση με άλλα πιο μολυντικά καύσιμα. Αλλά βεβαίως αυτό δεν θα πρέπει να αποβεί σε ζημία το, της ε, προώθησης ε, των, των εναλλακτικών μορφών ενέργειας. Ε, επίσης θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι το μεθάνιο συμβάλλει πολύ περισσότερο σε την δημιουργία αερίων του θερμοκηπίου και επομένως θα πρέπει οπωσδήποτε να προωθηθεί η έρευνα έτσι ώστε να απαλληλθεί η η ε, ε, επικινδυνότητα της ε, διάθεσης του μεθανίου στον αέρα. Βεβαίως αυτό δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσης εργασίας, το είπα και προηγουμένως. Εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι ο εισηγητής έχει λάβει υπόψη πολλά στοιχεία και από άλλες πολιτικές ομάδες και αυτό είναι θετικό. Ευχαριστώ κύριο Στοσενόφσκι, εξ ονόματος του ECR. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Γιώργ για το πρώτο αυτό προσχέδιο έκθεσης. Είναι μια εξαιρετική αφετηρία για τις συζητήσεις που θα έχουμε. Επίσης, συμφωνώ με αυτό που είπε και εκείνος εισηγητικά. Όπως είπε, κατέβαλε προσπάθεια προκειμένου η έκθεση αυτή να αφορά πραγματικά το υγροποιημένο φυσικό αέριο και να περιλαμβάνει η έκθεσή του τα σημαντικότερα ζητήματα σε σχέση με το LNG και να μην άπτεται η έκθεσή του διαφόρων άλλων θεμάτων που απασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς λοιπόν από την πλευρά μας θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να μην μπερδέψουμε τα θέματα. Συμφωνώ με τον συνάδελφο Γιώργ ότι στόχος μας σε αυτή την έκθεση είναι να μην φτιάξουμε μια έκθεση χριστουγεννιάτικο δέντρο η οποία θα άπτεται πολλών και διαφόρων θεμάτων, αλλά να επικεντρωθούμε σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα του υγροποιημένου φυσικού αερίου. Είναι πολύ σημαντική η πρόσβαση σε όλη την Ευρώπη ε, προς αυτό το LNG. Δεν θα πρέπει πρόσβαση σε αυτό το ε, υγροποιημένο φυσικό αέριο να έχουν μόνο κάποιοι συγκεκριμένοι, αλλά να αποτελέσει έναν βασικό πυλώνα της ενωσιακής πολιτικής μας το υγροποιημένου φυσικού αερίου, προκειμένου να εξασφαλίζεται και η ασφάλεια εφοδιασμού. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό και για τη σταθερότητα του συστήματος μας. Χρειαζόμαστε λοιπόν πολλά σημεία πρόσβασης, κάτι που μας προσφέρει το υγροποιημένο φυσικό αέριο, γιατί μέσω αυτού αποκτούμε την επιδιωκόμενη από εμάς ανεξαρτησία στον τομέα της ενέργειας. Από αυτή την άποψη λοιπόν θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον εισηγητή για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε μέχρι στιγμής και θεωρώ ότι ο ίδιος έχει επιδείξει μια εξαιρετική στάση σε όλη αυτή τη διαδικασία. Πρόεδρος, εκ μέρους της Άλντε, η κυρία Καρολίνα Πούντσετ, που εδώ και τρεις μήνες είναι πλήρες μέλος της, ε, τακτικό μέλος της ε, Επιτροπής μας. Πρώτα απ' όλα, όπως και οι υπόλοιποι σκιώδεις, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γιούρκο για την επικοδομητική του ε, στάση και για τη διάθεσή του να συμπεριλάβει όλα τα πολλά και διαφορετικά σημεία. και τουλάχιστον το έκανε αυτό με τα σημεία της Άλντε. Πρώτα απ' όλα, θέλω να σας πω ότι μου φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερο σημαντικό να ε, υπάρξει μεγάλη συμφωνία σχετικά με την, ε, με το ισχυρό μήνυμα το οποίο θα πρέπει να σταλεί στην Κομισιόν έτσι ώστε να μην επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος ε, που ε, κόστησαν πολλά χρήματα σε δημόσιες επενδύσεις οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται και δεν αποδίδουν καθόλου. Αυτό είναι σημαντικό να σταλεί ως μήνυμα στην Κομισιόν. Επίσης οι προβλέψεις κατανάλωσης να γίνονται με τρόπο ανεξάρτητο από ανεξάρτητες αρχές αρχές γιατί νομίζω ότι αυτό άλλωστε απασχολεί όλες τις πολιτικές ομάδες. Επίσης, θεωρώ ότι είναι εξίσου σημαντικό, όπως έλεγε ο κ. Ζανονέτη προηγουμένως, ε, ε, να μην παρεμποδιστεί από το αέριο, από το φυσικό αέριο, ε, η, η χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πάντα υπό το φως των αναγκών καταπολέμησης των συνθήκων που οδηγούν στην κλιματική κλιματική αλλαγή. Βεβαίως ακόμα δεν υπάρχει συμφωνία, ωστόσο η ομάδα μας θα συνεχίσει να εργάζεται έτσι ώστε να προκύψει συμφωνία, γιατί υπάρχει το ζήτημα των εκπομπών ε, μεθανίου που αναφέρθηκε άλλωστε και από τον ε, σύντροφο της σοσιαλιστικής ομάδας. Πρόκειται ε, για ένα πάρα πολύ σημαντικό ε, ζήτημα. Ε, οι εκπομπές μεθανίου που είναι 80 φορές πιο επικίνδυνες από τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακος είναι ένα θέμα ιδιαίτερα επικίνδυνο, σημαντικό για όλες τις χώρες γιατί συμβάλλουν ιδιαίτερο στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Εμάς μας ενδιαφέρει βεβαίως ε, η ε, σωστή χρήση της ξυλίας. Μας ενδιαφέρει να διατηρηθεί η βιωσιμότητα ε, των δασών από τα οποία κόβεται αυτή η ξυλία. Αυτό που θέλουμε είναι στο μέτρο του δυνατού να χρησιμοποιούνται καθαρές μορφές οι οποίες θα αποφεύγουν την υπερβολική ε, προ, έκκληση συγγνώμη, αερίων ε, μεθανίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Από τους ε, πρασίνους, ο συνάδελφος Γιάκοπ Νταλούντε, που αντικαθιστά το κύριο Έριξον. Πήρε τη θέση του πριν από μερικές εβδομάδες, επίσης από τη Σουηδία, από ό,τι ξέρω. Και ο συνάδελφό μα αυτό είναι ακόμα ένα μέλο ε, τη ειδική κυβέρνηση που προέρχεται από την Επιτροπή μας. Πόσα τέτοια μέλη ευρωπαϊκών κυβερνήσεων πέρασαν από εδώ. Χάνουμε τους συναδέλφους μας ε, <laughs> για να πάνε στις κυβερνήσεις. Και εσάς, συνάδελφε, το μέλος σας μάλλον στη ειδική κυβέρνηση θα είναι. Το ελπίζω, λέει ο μιλητής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον εισηγητή που σημείωσε κάποια πρόοδο στην έκθεση, παρότι από τη δική μα σκοπιά πολλά μένουν ακόμα να γίνουν. Τέσσερι παρατηρήσεις. Πρώτον, αυτή η στρατηγική δεν πρέπει να ε, υφίσταται εν κενό, αλλά σε ένα πλαίσιο. Και αυτό το πλαίσιο είναι οι προτεραιότητες ε, της Ευρωπαϊκή Ένωση για το κλίμα και την ενέργεια. Πρέπει λοιπόν ε, να επικεντρωθούμε στην μείωση της ζήτησης, στην ενεργειακή απόδοση και τη ΑΠΕ, καθώ και μία στρατηγική εξόδου για το φυσικό αέριο. Θα πρέπει λοιπόν να ιεραρχήσουμε ως προτεραιότητα αυτή την πολιτική και για τις ε, επενδύσεις ε, ως προς τις υποδομές. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τις υφιστάμενες ε, τάσεις ως προς τη ζήτηση φυσικού αερίου. Τα ισχύοντα σχέδια για τα μελλοντικά έργα βασίζονται σε προσβλέψεις για αύξηση της ζήτησης. Όμω αυτή τη στιγμή πέφτει η ζήτηση φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Με τη σημερινή μας ικανότητα εισαγωγή μπορούμε να καλύψουμε πάνω από 50% των αναγκών. Ενώ μάλιστα γίνεται και ελλειπή μερική αξιοποίηση των υποδομών. Και χάρη στην ενεργειακή απόδοση και τις ε, πολιτικές ε, ΑΠΕ ε, με την υλοποίηση των στόχων του 2030, κατά ψευθενότητα θα συνεχιστεί αυτή η φθήνουσα τάση ζήτηση για το ψυχοαέριο. αέριο. Αυτό θα πρέπει να ενσωματωθεί στην έκθεση. Μετά, χρειαζόμαστε βελτιωμένη ανάλυση της ζήτησης όπως έχει ήδη ζητηθεί από το Ελληνικό Συνέδριο και από πολλές μελέτες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει με προσοχή να αναθεωρήσει την ανάλυση της για τη ζήτηση φυσικού αερίου και την αξιολόγηση κινδύνων ε, και δυνατοτήτων βάσει των πραγματικών ε, δεδομένων που μπορούμε να βρούμε για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και χρειαζόμαστε καλύτερη ορολογία για το methane leakage, τη διαρροή μεθανίου. Βλέπουμε λοιπόν μεγάλες φθενότητες μεθανίου ε, και αυτό έχει πολύ σημαντικό αντίκτυπο σε ό,τι αφορά την ε, αύξηση της, ε, προθε... της θερμοκρασίας του πλανήτη, της υπερθέρμανσης του πλανήτη και δεν μπορούμε λοιπόν πλέον να θεωρούμε το φυσικό αέριο ως πηγή ενέργειας χαμηλού, χαμηλών εκπομπών βλέπουμε ότι σε άλλες περιοχές του κόσμου υπάρχει ε, σημαντική εξάρτηση από την υδρογμάτωση, το fracking. Γι' αυτό και εμείς θα πρέπει να επικεντρωθούμε ε, σε περαιτέρω μελέτες για τις ε, επαρκείς, ε, ακριβείς μάλλον, επιπτώσεις της ενέργειας και σε ό,τι φορά τις εκπομπές διευθυντήτου του άνθρακα. Σας ευχαριστώ. Θέλει κανείς άλλος να πάρει το λόγο. Η κυρία Μπερμέχο, παρακαλώ. Of, από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη εξ ονόματος του κυρίου, του συναδέλφου ε, νεοκλειή, ο οποίο δυστυχώ δεν μπορεί να είναι. Δεν είναι δυνατόν να είναι εδώ. Δεν είναι δυνατόν να, αφήσουμε, να αφήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο λιγοπόλιο του ε, αερίου την ενεργειακή πολιτική, γιατί δεν του ενδιαφέρει το γενικό συμφέρον. Ε, υπάρχουν και άλλε δυνατότητε συμβατικών μέτρων, όπω στην Κύπρο. Αλλά έχουμε δει ότι, ας πούμε, σε χώρες όπως η Ισπανία, το αέριο έχει γίνει ή ε, ο παράδεισος των καταχραστών. Ε, μπορώ να σας πω ότι υπάρχουν ας πούμε πάρα πολλές εγκαταστάσεις οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται καθόλου ή υποχρησιμοποιούνται και εντωμεταξύ φουσκώνουν τις ε, ε, τους λογαριασμούς. Ε, επίσης, εταιρείε όπως η Καστόρ, η οποία ε, καταστρατηγεί όλες τις περιβαλλοντικές αξίες και όλους τους περιβαλλοντικούς νόμους, γιατί δεν ενδιαφέρεται για τον τρόπο με τον οποίο παράγεται το υγροποιημένο αυτό αέριο. Επίσης, αναφερθήκαμε ήδη εις την δυνατότητα την δημοκρατική και με κυρίαρχο τρόπο Απόφαση των λαών. Ε, οι λαοί μπορούν να αποφασίσουν να μην δέχονται τέτοιου είδους, ε, ε, να μην δέχονται προϊόντα τα οποία προέρχονται από μη οικολογικέ διαδικασίες όπως ας πούμε είναι η υδρορογμάτωση. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Βέρα. Θα τα πω στη γλώσσα μου, λέει η κυρία Πιλάρ Καστίγιο. Ε, πιστεύω ότι ο σλένφος Ανδρέας Γιούρκ ε, ε, δούλεψε πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι άλλωστε ε, και οι σκιώδεις αναγνώρισαν την καλή αυτή εργασία. Ε, στην αρχή της παρέμβασής του είπε ε, κάτι το οποίο υπογράμμισε και μετά και το οποίο μου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή ότι θα πρέπει να είναι ισορροπημένη και καλά εστιασμένη η έκθεση αυτή. Βεβαίως αυτή η αρχή ισχύει για όλες τις εκθέσεις, αλλά εδώ νομίζω ότι ισχύει ακόμα περισσότερο, γιατί όπως είπε και ο εισηγητής, ε, το θέμα αυτό δεν θα μπορεί να είναι μία έκθεση όπου ο καθένας θα βάλει το μακρύ του και το κοντό του, δεν μπορεί να γίνει χριστουγεννιάτικο δέντρο, γιατί διαφορετικά ε, σε μια τέτοια περίπτωση θα χανόταν ε, η ε, ουσία της έκθεσης. Ξέρουμε ότι αυτό αυτό έχει ε, χρησιμοποιηθεί, ε, μάλλον έχει συμβεί πάρα πολλές φορές, ε, δηλαδή δημιουργούνται εκθέσεις και ζητήματα τα οποία είναι τόσο μεγάλα και περιλαμβάνουν τόσα πολλά πράγματα που χάνεται η ουσία και δεν μπορούν να την πιάσουν την ουσία αυτή και οι πολίτες. Το θέμα της, του υγροποιημένου αερίου και της παροχής του υγροποιημένου αυτού αερίου είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για γιατί μπορεί να μειώσει την εξάρτηση ε, από αυτήν την ε, αποκλειστική και μεγάλη εξάρτηση που ε, έχουν πάρα πολλές χώρες από το φυσικό αέριο, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σπάει λοιπόν η δυνατότητα παροχής υγροποιημένου αερίου την, την κατάσταση που αντιμετωπίζουν πολλές χώρες. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο θέματα. Πρώτον, ότι το ζήτημα αυτό συνδέεται άμεσα και άλλωστε αυτό καταδεικνύεται και από κάποιες από τις υποβληθήσεις τροπολογίες Δηλαδή αναφέρομαι στην ε, ε, υπογράμμιση της ε, σημασίας των διασυνδέσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί διαφορετικά όλο αυτό το σύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει και ο στόχος της διαφοροποίησης της προμήθειας και της παροχής δεν θα μπορούσε να ικανοποιηθεί. Και κάτι άλλο το οποίο ανέφερε και ο Σένφος Μπούζεκ, ε, δηλαδή ότι θα πρέπει να βελτιωθεί ε, όσο ε, γίνεται περισσότερο, να γίνει όσο, όσο καλύτερη γίνεται η χρήση των υπαρχουσών δομών και θα πρέπει να επιμείνουμε στην έκθεση αυτή να ε, υπογραμμιστεί η σημασία και η χρήση των ήδη υφισταμένων δομών ε, γιατί με τον τρόπο αυτό θα έχουμε μια, έναν καλό υπολογισμό κόστους κόστους-οφέλους και δεν θα δημιουργήσουμε ανώφελες νέες υποδομές. Δεν θέλω τίποτα άλλο να πω. Νομίζω ότι ε, εδώ έχουμε μια πολύ σημαντική έκθεση, καλά εστιασμένη η οποία έχει σαν κύριο μέλημα την διαφοροποίηση της ενέργειας αλλά και την ασφάλεια της παροχής ενέργειας και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας. Κύριε Συγγνώ... κύριος, συγγνώμη αν ε, δεν προφέρω σωστά το όνομά σας. Ευχαριστώ κύριε Μπούζεκ, αγαπητά μέλη της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ για την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε σε αυτό το θέμα. με μια σειρά από μέλη της Επιτροπής σας και με τους κοιόδης συζητητές. Συμφωνούμε απολύτως με, τις βασικές, με τα βασικά συμπεράσματα της ε, έκθεσής σας. Θα τα λάβουμε υπόψη την ε, διαφοροποίηση και την ανάγκη διαφοροποίησης προκειμένου να βελτιωθεί η ενεργειακή ασφάλεια και η ασφάλεια εφοδιασμού στην Ευρώπη. Όπως είπαν πολλοί και από εσάς, είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξευρεθεί η σωστή ε, ισορροπία η βιωσιμότητα, θα πρέπει να εξετάσουμε το LNG και ολόκληρο το θεματολόγιο για, την, ε, ε, για το φυσικό αέριο με βάση τους στόχους για το κλίμα και την ενέργεια. Προσπαθούμε να συνδυάσουμε και να προσαρμόσουμε την στρατηγική μας και την πολιτική μας ε, και εν ώψη των στόχων για το 2030 και 2050 πράγματι η ζήτηση θα μειωθεί. Αυτό που έχουμε διαπιστώσει είναι ότι καθώς ε, μειώνονται οι εισαγωγές, θα, καθώς μάλλον μειώνεται η εσωτερική ε, παραγωγή, ε, η ζήτηση θα διατηρηθεί σε σχετικά σταθερά επίπεδα. Γι' αυτό δεν θα μπορέσουμε να αποφύγουμε τις σημαντικές, εδώ που τα λέμε, εισαγωγές φυσικού αερίου στο μέλλον. Πρέπει λοιπόν να πω ότι το LNG δεν είναι εμπόδιο στις ΑΠΕ, Αντιθέτως, ε, είναι ε, μια, ένα συμπληρωματικό στοιχείο στο ενεργειακό μείγμα μας. Είναι ένα καύσιμο χαμηλών εκπομπών ε, άνθρακα συγκριτικά. θα πρέπει λοιπόν να αξιοποιηθεί πλήρως στο μελλοντικό μας ενεργειακό μείγμα και θα πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε και με άλλους εταίρους σε ολόκληρο τον κόσμο και με βιομηχανίες και εταιρείες που συμμερίζονται τους δικούς μας στόχους. Όσον αφορά την ενιαία αγορά, όπως υπόθηκε, είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλιστεί η προσιτότητα ε, και η προσβασιμότητα. Εμείς δεν θέλουμε παρά τις ελάχιστες αναγκαίες επενδύσεις προκειμένου να υπάρξει αυτή η διασύνδεση και ιδίως από την άποψη ότι μακροπρόθεσμα πράγματι η ζήτηση σε φυσικό αέριο θα μειωθεί και λόγω της ε, ενεργειακής αποδοτικότητας. Οπότε αυτή τη στιγμή δεν θα ήταν σωστό να υπάρξουν τεράστιες επενδύσεις στο LNG σε κάθε κράτος μέλος, αλλά θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι πραγματικά αναγκαίες επενδύσεις προκειμένου όλα τα κράτη-μέλη να έχουν πρόσβαση στο LNG και, στην, ε, και στα αποθέματα. Σε διεθνές επίπεδο θα πρέπει να συνεργαστούμε με τους εταίρους μας και όσον αφορά το θεματολόγιο για τη βιωσιμότητα, είπα την Αυστραλία, αλλά και άλλους πολύ σημαντικούς εταίρους στις χώρες του κόλπου και, την, και στην Αφρική οι οποίες θα είναι και εκείνες οι οποίες θα μας ε, προμηθεύουν κατά κύριο λόγο με το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Θα ήθελα λοιπόν τελειώνοντας να σας ξαναευχαριστήσω για όλη τη συνεργασία που είχαμε στο θέμα αυτό και ανυπομονώ να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας και να καλέσω βεβαίως και από τη δική μου πλευρά να, τα κράτη-μέλη να κάνουν ό,τι χρειάζεται προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτή η διασύνδεση της ε, ενιαίας ε, αγοράς ενέργειας. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο κύριος Πρόεδρος, για την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτήν την παρουσίασή της. Δεν θέλετε και πολλές επενδύσεις από ό,τι μας είπατε, αν κατάλαβα σωστά. Ωραία. Κύριε Σιγητά, Κύριε Άντρα Γιούρ, ποια είναι η δική σα γνώμη για όλα αυτά που ακούστηκαν. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις πολύτιμες παρατηρήσεις τους και στη βάση των όσων ακούσαμε σήμερα αλλά και ε, στη βάση των ε, συναντήσεων σκιωδών που είχαμε μέχρι στιγμή, είμαι πολύ αισιόδοξο ότι θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε έναν καλό συμβιβασμό και όπως είπα και νωρίτερα είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει η ευρύτερη δυνατή ε, συμφωνία. Γιατί αν καταφέρουμε να μιλήσουμε με μία φωνή, θα καταφέρουμε να επηρεάσουμε τα πράγματα σε αυτόν τον πολύ σημαντικό για το μέλλον τομέα της ενεργειακής πολιτικής. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε για την έκθεσή σου, για την παρουσίασή σου και όλους εσάς αγαπητοί συνάδελφοι για τις συζητήσεις που έγιναν. Βεβαίως να ευχαριστήσω και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αύριο το πρωί, στις 9 το πρωί, συντονιστές όσοι είστε τυχεροί να είστε, 10 η ώρα ψηφοφορίε. Οπότε θα τα πούμε ε, με όλους στις 10, με τους συντονιστές σε 9 το πρωί. Ευχαριστώ πολύ, θα τα πούμε αύριο. Γεια σας.